Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώ ήρθατε θερμά στη συνεδρίασή μα την πρωινή σήμερα. Έχουμε πολλές ψηφοφορίες που προβλέπονται στην ημερήσια διάταξη και προτού περάσουμε στην ημερήσια διάταξη επιτρέψτε μου μια ομάδα επισκεπτών από την Καλαβρία να καλωσορίσω που από τον συνάδελφο Πύλο έχουν προσκληθεί. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος εσείς ε, επισκέπτες από την Καλαβρία. Και περνάμε τώρα στη συνέχεια στο σημείο 22 της ημερήσιας διάταξης. Convention, σύμβαση και διεθνές εμπόριο των απειλούμενων με εξάλληψη αγρίων ζώων, πανίδας και χλωρίδας, σάιτης. Έχετε όλοι τις κάρτες για την ψηφοφορία σας επειδή ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας. Παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες που έχετε. So, Εντάξει, λοιπόν ξεκινάμε κιόλας. Έχουμε την τροπολογία 28 με προφορική, προφορική τροποποίηση. Ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ, εσείς έχετε τον λόγο. Είναι κατά της προφορικής τροποποίησης η ομάδα μου. Οι πράσινοι είναι κατά της προφορικής τροποποίησης. Επίση Επίσης οι φιλελεύθεροι. Έτσι λοιπόν δεν θεωρείται αποδεκτή η προφορική τροποποίηση. Ψηφίζουμε την τροπολογία 28 ως είχε στην αρχική μορφή της. Τώρα θα πρότεινα όμως συνάδελφοι να ψηφίζουμε σηκώνοντα το χέρι και μόνο αν υπάρχει κάποια αμφιβολία ηλεκτρονικά. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ να σηκώσουν το χέρι υπέρ 28 στην αρχική της διατύπωση. Ευχαριστώ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Περνάμε τώρα στην 27, τροπολογία 27. Ποιοι είναι υπέρ της 27. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Περνάμε στην 29, τροπολογία 29. Ποιοι είναι υπέρ της 29. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τώρα η 30. Με προφορική τροποποίηση. Είμαστε κατά αυτών των δύο προφορικών τροποποιήσεων. Είσαστε κατά και των δύο. Λοιπόν, 30 και 31 εννοείται αυτές τις δύο, έτσι οι προφορικές τροποποίησεις. Ψηφίζουμε στην αρχική διατύπωση. Ποιοι είναι υπέρ της 30 στην αρχική της διατύπωση. Κατά της 30. Απορρίφθηκε. Περνάμε στην 31 τώρα. Χωρίς προφορική τροποποίηση. Ποιοι είναι υπέρ της 31. Κατά και αυτή απορρίφθηκε. 32. Έχει αποσυρθεί όμως η 32. Περνάμε τώρα. Η 33 και αυτή έχει αποσυρθεί. Και έτσι περνάμε στην τροπολογία 34. Ποιοι είναι υπέρ τη 34. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 35. Υπέρ τη 35 παρακαλώ κατά αποχές εγκρίθηκε 36 αποσύρθηκε η 36 και έχουμε την 38 και την 54 που είναι ταυτόσιμες μπορούμε να τις ψηφίσουμε από κοινού ποιοι είναι υπέρ της 38 και υπέρ της 54 κατά αποχές εγκρίθηκαν 39 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά ψηφίζουμε ποιοι είναι υπέρ της 39 άρχεται η ψηφοφορία εννοώ Ευχαριστώ. Πέρας ψηφοφορίας. Ήταν καλό το ότι ψηφίσαμε. 25 υπέρ, 24 εναντίον, μία αποχή. Ήταν πολύ στενή η διαφορά λοιπόν πράγματι. 40. Ποιοι είναι υπέρ τη 40. Παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Το ίδιο αποτέλεσμα υποθέτω, αλλά θα ελέγξουμε και πάλι ηλεκτρονικά. 40 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Μάλιστα. Το αντίστροφο αποτέλεσμα. 25 υπέρ 26 εναντίον. Καμία αποχή. Απορρίφθηκε λοιπόν η 40. 41 τώρα. Ποιοι είναι υπέρ της 41. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 41. Πέρας ψηφοφορίας. 25 υπέρ, 26 εναντίον. Απορρίφθηκε. 42 τώρα. Υπέρ τη 42. Κατά. Θα κάνουμε πάλι το ίδιο. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τη 42. Πέρας ψηφοφορίας. Μάλιστα. Όλο και βελτιώνεται η κατάσταση. 25 υπέρ, 25 εναντίον, ισοψηφία απορρίπτεται. Δεν λειτουργήσε η συσκευή μου, Πρόεδρε. Ε, τότε να καθίσετε κάπου αλλού για την επόμενη ψηφοφορία, τις επόμενες ψηφοφορίες. Αλλάξτε θέση. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, αν είναι εντάξει, νομίζω ότι θα έπρεπε ομού σαν ομάδα ε, ε, να είχαμε ψηφίσει, να ψηφίσαμε τις τροπολογίες 54 ε, και 53 και ο ρόλος γι' αυτό είναι ότι όλες αφορούν διαφορετικά είδη στη Μαδαγασκάρη και υπάρχει πολύ μικρή απόκληση απόψεων για αυτό το θέμα έχουμε ευθυγραμμιστεί για το site που πρέπει να εγκριθεί δηλαδή τουλάχιστον από πλευρά site για αυτά τα είδη και ουσιαστικά μπορεί να υπάρχουν λόγοι να ενταχθούν αλλά όχι ακόμα τα επιστημονικά τεκμήρια και δεν θα είχε νόημα να υπάρξουν αναείδος διότι δεν υπάρχει κάποια διαφορά και από την ίδια τη Μαδαγασκάρη προτάθηκαν να ενταχθούν στις δεν ξέρω αν Κρήτο αν θέλετε να τοποθετείτε εσείς. Δεν, λυπάμαι, δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Ψηφίζουμε τη 42 ακόμα. Είπε η συνάδελφος μόλις πριν ότι δεν λειτουργούσε η συσκευή της. Επειδή ήταν ισοψηφία το αποτέλεσμα 25-25 στις ψήφους, από πλευράς γραμματείας μου είπαν ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας παραμένει ως έχει, δεν μπορεί να αλλάξει τέρμα. Έχουμε όμως ένα πρόβλημα, ότι δεν έχει ένα μέλος την κάρτα του για να ψηφίζει. Also in der Geschäftsordnung steht im Zweifel λέει ο κανονισμός αν υπάρχει αμφιβολία θα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Όποιος δεν μπορεί να ψηφίσει ηλεκτρονικά επειδή δεν έχει κάρτα τότε ε, και θα έρθει ο τεχνικός σε εσά κυρία για να ε, επισκευάσει τη συσκευή σας. Ίσως μπορείτε να αλλάξετε θέση για τις επόμενες ψηφοφορίες για να μην υπάρξει πρόβλημα. Απορρίφθηκε 42. Συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε στην άλλη περίπτωση. 43 τώρα. Υπέρ της 43. Παρακαλώ. Κατά. αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 43, άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. 26 υπέρ, 26 εναντίον. Απορρίφθηκε. 44. Υπέρ της 44 παρακαλώ. κατά. Ίδια διαδικασία λοιπόν πάλι. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 44. Πέρας ψηφοφορίας. υπέρ, 26 εναντίον απορρίφθηκε. Τροπολογία 45 υπέρ κατά θα ελέγξουμε και πάλι ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 45 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας 26 υπέρ, 27 εναντίον και αυτή απορρίφθηκε. Περνάμε στις 46 τώρα. Με προφορική τροποποίηση. Δεν υπάρχει αντίρρηση για αυτήν την προφορική τροποποίηση. Υπέρ τη 46 παρακαλώ. Κατά. Εγκρίθηκε. Ε, τότε να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε τις 46 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Λοιπόν, είχα δίκιο. 33 υπέρ, 20 εναντίον, μία αποχή, εγκρίθηκε η 46. 47 τώρα, με προφορική τροποποίηση, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 48 υπέρ, υπέρ της 48 κατά άποχες πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας αποτέλεσμα 25 υπέρ 29 εναντίον απορρίφθηκε τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 50 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 51 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 52 υπέρ κατά αποχές και αυτή απορρίφθηκε 53 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε φτωχέ μου Κρήτον απορρίφθηκαν όλες σχεδόν όλες. 55. Τροπολογία 55 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στην 59. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 61 αποσύρθηκε 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε βελτιώνεται η κατάσταση τώρα Κρήτων 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μάλιστα να τα κάνουμε να ψηφίσουμε ομού όλες κατηγοριοποιημένες μαζί 68 όχι μέχρι την 68, όχι, αντίρρηση, εντάξει, λοιπόν. Που είμαστε στην 64, υπέρ λοιπόν της 64, κατά αποχές εγκρίθηκε, 65 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε, 66 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε, 67 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε, 68 υπέρ, κατά Απόχες. Εγκρίθηκε. Λοιπόν, περνάμε τώρα στις αιτιολογικές σκέψεις. 1. Υπέρ. Κατά. Απόχες. 2. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίφθηκε. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 4. Υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 5 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε σχεδόν ταυτόσιμη λέει εδώ είναι η 6 και η 7 λοιπόν από κοινού θα τις ψηφίσουμε 6 και 7 υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν Οκτώ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε έντεκα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 12 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συγγνώμη τώρα που πάμε τώρα πάμε στην προφορικέ στις προφορικές τροποποίησεις στο ΙΑ δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση κατά της προφορικής τροποποίησης. Θα ψηφίσουμε λοιπόν ποιοι είναι υπέρ της προφορικής τροποποίησης στο ΙΑ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 17 με προφορική τροποποίηση. Ναι, συνεχίζουμε. 18. Εντάξει, σωστό. Ψηφίζουμε την 18. Πάει η 17, έχει διευθετηθεί ήδη. 18 υπέρ, λοιπόν. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 20 υπέρ. 21 πρώτα λέγεται στον πρόεδρο. Ναι, 21 υπέρ, συγγνώμη. Κατά αποχές εγκρίθηκε. «23. Σε τμήματα η ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ». «Κατά» αποχές εγκρίθηκε το πρώτο τμήμα. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της 23. Ένα Ένας από το ΕΛΚ είναι παραπάνω από τις ψήφους από τα μέλη του ΕΛΚ. Κάποιος να μην ψηφίζει, να μην συμμετέχει λοιπόν. Έχετε έναν παραπάνω από το ΕΛΚ. Συντονιστή, τι λέτε. Εντάξει. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας τώρα. Ωραία. 33 υπέρ, 23 εναντίον. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα της 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 24 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία ποιοι είναι υπέρ του ψηφίσματος θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά ηλεκτρονικά λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά Πέρας πληροφορία. Μάλιστα. Σαφές το αποτέλεσμα. 48 υπέρ, 2 εναντίον, 6 αποχές. Συγχαρητήρια. Θερμά συγχαρητήρια στους συντάκτες για αυτή την πολύ σημαντική έκθεση. Ευχαριστώ λοιπόν. Και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερησία διάταξη, το 23. Ασφάλεια του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Η είναι ο συνάδελφος Μπόγκουσλαβ Σόνικ. Περνάμε αμέσως στην ψηφοφορία και ψηφίζουμε. Τροπολογία 3. Uh, Αρχίζουμε λοιπόν. Τροπολογία 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38. υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6, που είναι συμβατή με την προηγούμενη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 39, κατά τμήματα ψηφοφορία, πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στην τροπολογία 44 Ψηφίζουμε μόνο για το υπόλοιπο τμήμα που περιγράφεται εδώ στο κείμενο. Ποιος είναι υπέρ αυτού του τμήματος. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, δεν είναι ξεκάθαρο. Για το δεύτερο τμήμα να ψηφίσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ποιο είναι... Ψηφίζουμε για το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. 31 ψήφοι υπέρ, 25 κατά. Εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 45 καταπίπτει. Τροπολογία 46, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 48, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να την ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. 26 ψήφοι υπέρ, 30 ψήφοι κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 και 52 είναι ταυτόσιμες. Σας ψηφίσουμε μαζί. ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 15 καταπίρτη. Στη 16 ψηφίζουμε μόνο για το υπόλοιπο τμήμα του κειμένου που μένει. Ποιος είναι υπέρ λοιπόν αυτού του υπολείπου, υπέρ για τη 16. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Α, έφτασε και η κάρτα της ψηφοφορίας σας επιτέλους. Λήξη της ψηφοφορίας. 36 υπέρ, 20 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. Η 55 καταπίπτει. Και η 54 καταπίπτει. Και στην τροπολογία 17 ψηφίζουμε για το υπόλοιπο κομμάτι που έχει απομείνει ψήφι υπέρ της 17 για το υπόλοιπο κομμάτι που έχει απομείνει. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 56 καταπίπτει. Και η 18 καταπίπτει. Τροπολογία 19. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 57 καταπίπτει. Ψηφίζουμε την 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 58 καταπίπτει. 59 υπέρ. Υπέρ πάλι για την 59. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. Ε, συγγνώμη, απορρίπτεται. Τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για τις αιτιολογικές σκέψεις και παραθέσεις, τροπολογία 23 του κ. Ούλμερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα για το σύνολο της έκθεσης. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. 52 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά και 4 αποχές. Εγκρίνεται η έκθεση. Συγχαρητήρια στον συνάδελφο κύριο Σόνικ. Ελπίζουμε επιτέλους να υπάρχει ασφάλεια του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο και να μην συμβεί ποτέ ξανά τίποτα. Και περνάμε στο σημείο 24, πολιτική ποιότητα των γεωργικών προϊόντων, τι στρατηγική πρέπει να ακολουθήσουμε. Η η Πιλάρα Γιούσο. Ψηφίζουμε τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Εντάξει, θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 5. Πέρας ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 32 εναντίον. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. Μα ήταν σαφέστατο το αποτέλεσμα. Δύο τρίτα, ένα τρίτο ήταν. Τοπολογία τέσσερις τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τοπολογία επτά υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Στην 8 έχουμε σε τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 9 σε τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 11 σε τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 13 δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε πάει αυτή είναι γλωσσικό θέμα 14 τώρα υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά ψηφίζουμε τη 14 πέρας ψηφοφορίας ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Κάποιος πρέπει να αφαιρέσει την κάρτα του, να μην συμμετέχει. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ λέω. Τώρα εντάξει. Πέρας ψηφοφορία λοιπόν. Μάλιστα, αυτό είναι αποτέλεσμα. Είναι συντριπτική πλειοψηφία λοιπόν. 56 υπέρ. Ένας εναντίον. Μάλιστα, εγκρίθηκε. 15 τώρα υπέρ. κατά αποχές απορρίφθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν, έστω ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. 36 υπέρ, 20 εναντίον παρατηρώ, βλέπω ότι οι κινήσεις των χεριών σας δεν είναι σαφείς πλέον. Λοιπόν, εγκρίθηκε η 15, 16 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε και ψηφίζουμε τώρα σε τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 51 υπέρ, 5 εναντίον, μία αποχή. Θερμά συγχαρητήρια Πιλάρα Γιούσο για αυτή τη γνωμοδότηση που συντάξατε. Θερμά συγχαρητήρια. Και περνάμε στο επόμενο σημείο που θα ψηφίσουμε του Μάριο Πυρίλο. επενδυτικά σχέδια σε ενεργειακή υποδομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Εισηγητής ο κύριο Πυρίλο, είπαμε. Περνάμε ήδη στην τροπολογία 2 του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 14 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 15 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 16 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 17 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 18 υπέρ κατά αποχές νομίζω εγκρίθηκε αυτό θα έλεγα θα ελέγξουμε ωραία άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά 18 ψηφίζουμε τη 18 πέρας ψηφοφορίας Μάλιστα, σαφές το αποτέλεσμα. 34 υπέρ, 19 εναντίον, 4 αποχές. Εγκρίθηκε η 6 τώρα. Αποσύρθηκε η 6. Περνάμε στη 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 7. Υπέρ. Κατά Θα πρέπει να ελέγξουμε εδώ. Ψηφίζουμε την επτά άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Μάλιστα, αποτέλεσμα 23 υπέρ, 31 εναντίον, 2 αποχές, απορρίφθηκε, 8 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Κουραστήκατε όλοι. Δεν μπορώ να δω ποιο είναι το αποτέλεσμα. Αν ψηφίζουν ενωμένε οι ομάδε και τι γίνεται. Πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 8 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Ναι, είναι σαφές με το αποτέλεσμα αλλά δεν μπορούσα να το δω πιο πριν. 20 υπέρ 31 εναντίον, δύο αποχε απορρίφθηκε. Και ολοκληρώνουμε σχεδόν. Περνάμε στην τροπολογία 1 για το σύνολο του κειμένου. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 9, υπέρ, κατά, Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 9. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. 16 38 εναντίον 2 αποχές, απορρίφθηκε. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 56 υπέρ, καμία ψήφος εναντίον, μία αποχή μόνο. Θερμά συγχαρητήρια στον Μάριο Πυρίλο για την έκθεση αυτή. Θερμά συγχαρητήρια. Και ισχύει το ότι στις ενεργειακές υποδομές στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές προωθούνται ένα βήμα παραπέρα. Ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνατε για να συντάξετε αυτήν την έκθεση κύριε Πυρίλο. Λοιπόν, έτσι συνάδελφοι περνάμε τώρα στο σημείο 26 στην ημερήσια διάταξη. Έχει σημαντική υπόθεση αυτό το θέμα. Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές. Η συγγήτρια η κυρία Ρενάτε Ζόμερ. Και είχαμε προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών την 9η Δεκεμβρίου. Πολλές τροπολογίες έχουν κατατεθεί. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην εισηγήτρια για να σχολιάσει. Παρακαλώ κυρία Ζόμερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επειδή είναι ένα ευρύτατο θέμα αυτό, στο οποίο υπάρχει θα έλεγα ομοθυμία, συνενετικό πλαίσιο. Θα περιμένω δύο λεπτά μέχρι να ησυχάσουν οι συνάδελφοι. Πρόεδρος, λοιπόν ησυχία. Ξέρω, είχαμε τόσες ψηφοφορίες, πρέπει να συζητήσετε κάποια θέματα, το καταλαβαίνω. Όμως παρόλα αυτά, ησυχία. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορείτε έξω να συζητήσετε. Υπάρχει πολλής χώρος εκτός εθούσης. Λοιπόν, ωραία. Τώρα νομίζω πάμε καλύτερα. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ξεκινάμε και πάλι, η κυρία Ζόμερ. Ευχαριστώ για το ότι δεν κατατέθηκαν υπερβολικά πολλές τροπολογίες όπως πριν από ένα εξάμεινο ή και παραπάνω πριν στην πρώτη έκθεση που είχαμε. Αυτό οφείλεται στο ότι τώρα για αυτή τη δεύτερη έκθεση που έχουμε μπροστά μας πολλές τροπολογίες έχουν ενταχθεί στο κείμενο πλέον από εκείνες που είχαν προταθεί στο παρελθόν. Παρόλα αυτά, βέβαια, υπάρχουν πολλές ιδέες από τους συναδέρφους που διατυπώνονται και προτείνονται στις τροπολογίες τους. Και θα ήθελα σε κάποια άρθρα να αναφερθώ, δεν είναι δυνατόν να αναφέρω βέβαια τα πάντα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το άρθρο 7. Πρόκειται για την αξιοπιστία και το σωστό πλαίσιο της ενημέρωσης από πλευράς πληροφοριών υπάρχει ομοφωνία ότι θέλουμε να αποφύγουμε οπωσδήποτε παραπλάνηση των καταναλωτών να αποφύγουμε οπωσδήποτε μια παραπλάνηση. Και αυτό ανταποκρίνεται σε αυτό που είχα προτείνει στην έκθεσή μου. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας λοιπόν. Είμαι πρόθυμη υπό κάποιους όρους ε, για ορισμούς όσον αφορά τα νητράτα και όσον αφορά την έκθεσή μου για αυτό το άρθρο είμαι πρόθυμη τον ορισμό να τον τροποποιήσω κάπως είναι και μια πρώτη ιδέα αυτή που είχα, και είχα προτείνει ούτως ή άλλως. Μια τροπολογία των συναδέφων Σλούτερ και Χάση για την απαγόρευση όσον αφορά την απεικόνηση φρούτων ε, ή την, ε, ε, των άλλων συστατικών ουσιών είναι το θέμα του ορισμού. Τι είναι μικρή ποσότητα και τι όχι. Θα πρέπει να το συζητήσουμε. Απαγόρευση της κατηγοριοποίησης γάλακτος ως νοπού φρέσκου γάλακτος όταν είναι διατηρήσιμο επί μεγάλο, μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για παράδειγμα 10 μέρες δεν είμαι υπέρ του να απαγορευτεί να πούμε ότι είναι φρέσκο γάλα αλλά κάπως θετικότερα να το διατυπώσουμε να πούμε είναι νοπό φρέσκο γάλα το οποίο μπορεί να διατηρηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη Γερμανία σε κάποιες περιφέρειες έχουμε αυτή τη λύση και οι καταναλωτές την κατανοούν πολύ καλά και την αποδέχονται. Τώρα αν είναι δυνατόν να έχουμε ένα ευρύτερο μητρό με απαγορευμένες ουσίες ε, και ορισμούς ε, όσον αφορά απαγορεύσεις, αν ένα τέτοιο μητρό πρέπει να υπάρξει, το θεωρώ πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Διότι οι άνθρωποι είναι πάντα πολύ επινοητικοί και έτσι θα μπορούσαν και να το παρακάμπτουν κάτι τέτοιο. Έτσι πρέπει λοιπόν αντίστοιχα να είμαστε προσεκτικοί. Στο άρθρο 9 αντίστοιχες αναφορές. Τι πρέπει να αναφέρεται σε σχέση με τρόφιμα και τι όχι. Θα ήθελα στους Ιταλούς συναδέλφους να απευθύνω παράκληση την δική του τροπολογία όσον αφορά την επισήμανση private labor να εξηγήσουν τι εννοούν και τι θέλουν να κάνουν με αυτό. Εγώ μέχρι σήμερα πίστευα πάντα ότι αυτή την τροπολογία δεν θα μπορούσα να την εγκρίνω, δεν θα έπρεπε να την εγκρίνουμε. Ίσως όμως οι συνάδελφοι από την Ιταλία μπορούν να επεξηγήσουν ακριβώς εξειδικευμένα το αίτημά τους στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Μετά, όσον αφορά την διατηρησιμότητα μετά το άνοιγμα της ε, συσκευασίας, εντάξει, συμφωνώ, όμως αυτό το άρθρο πάει αρκετά μακριά, πολύ μακριά και δεν είναι ρεαλιστικό. Σε σχέση με την τροπολογία τώρα του συναδέφου Σλούτερ, επισήμανση, τικετοποίηση όσον αφορά τις διαστάσεις σε ποσοστά όπου εργασία παιδιών ή καταναγκαστική εργασία ή όταν εδώ το απαγόρευση του δικαιώματος του συνέρχεστε ε, είναι ε, στη ρίζα του, της παραγωγής. Κάτι τέτοιο δεν μπορώ να κατανοήσω πώς μπορεί να γίνει. Τώρα, για τις συζητήσεις που έπρεπε να γίνουν για τις τροπολογίες, για το άρθρο 9 παράδειγμα, για τις υποχρεωτικές ενδείξεις προέλευσης, δηλαδή αναφορά χώρας προέλευσης. Έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες που κατατέθηκαν σε σχέση με αυτό το άρθρο. Εγώ ίδια στην πρώτη μου έκθεση είχα προτείνει το κρέας σε, εκτός ε, του βοηού κρέατος που ρυθμίστηκε με την κρίση των ε, ε, βοηδών να προσέξουμε να μην υπάρχει παραπλάνηση όσον αφορά την χώρα προέλευσης. Εδώ υπάρχει επιθυμία προφανώς υποχρεωτικά το κρέας να επισημαίνεται, να ετικετοποιείται όσον αφορά την προέλευση του κρέατος. Θα μπορούσα να το δεχτώ αυτό. Είναι για το κρέας κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά για άλλα γεωργικά προϊόντα τώρα, σε αυτό τον κανονισμό, να πούμε ότι μια υποχρεωτική ένδειξη στην ετικετοποίηση για τη χώρα προέλευσης πρέπει να αναφέρεται, αυτό το θεωρώ αμφισβητήσιμο. Πρώτα απ' όλα για τα το φρέσκο κρέας, τα φρέσκα λαχανικά και τα νοπά φρούτα είχα καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Αλλά κατέληξα στο ότι είναι ίσως πιο, πιο ε, σκόπιμο να παραμείνουμε στις τομεακές ρυθμίσεις, διότι οι τομεακές αυτές διατάξεις και ρυθμίσεις μπορούν να είναι πιο ελαστικές και πιο εύκολα προσαρμόσιμες, ενώ διαφορετικά δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε στις ανάγκες. Παρακαλώ οι συνάδελφοι να προβληματιστούν και να το ξαναδούν. Μήπως έχει νόημα για τέτοιου είδους γεωργικά προϊόντα προϊόντα εκτός από το κρέας να έχουμε τις τομεακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν αντί να καθορίσουμε κάτι υποχρεωτικό σε αυτόν τον κανονισμό από πλευράς μας. Πιστεύω ότι πρέπει να έχει φυσικά τη δυνατότητα ο καταναλωτής από πού προέρχονται αυτά τα ε, προϊόντα ως πρώτη ύλη, ως προϊόντα αλλά πρέπει να είμαστε ελαστικοί, να μπορούμε να προσαρμοστούμε στις ανάγκες. Τώρα, για την ε, χώρα προέλευσης ε, η προέλευση των κύριων συστατικών ε, τροφίμων που αναφέρονται ως κυριότερα ή ουσιοδέστερα χαρακτηριστικά συστατικά στοιχεία ή σε μη επεξεργαστένα τρόφιμα όσον αφορά τα ουσιοδέστερα στοιχεία. Δύσκολο πρέπει να πούμε ότι είναι κάτι τέτοιο. Τα κανόνα μάλιστα ανέφικτο, αδύνατον διότι υπάρχουν και συστατικές ουσίες που αγοράζονται στην παγκόσμια αγορά και πώς μπορούμε να πούμε από πού προέρχονται. Η αγορά γίνεται ε, αυτών των προϊόντων ανάλογα με το από ποια χώρα είναι διαθέσιμα ή και από διαφορετικές χώρες κιόλα. Πώς μπορούμε όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο να το αναφέρουμε στην ετικέτα. Τεχνικά λοιπόν είναι ανέφικτο, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Για τη συνάδελφο Γιούτα, έχω το ερώτημα τι εννοεί με την ετικετοποίηση προέλευσης για τα τρόφιμα που αποτελούνται από μία συστατική ουσία. Τι είναι αυτό δεν θα είναι ε, νοπά ε, γεωργικά προϊόντα, αλλά πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό που στοχεύετε να κάνετε. Θα ήμουν ευγνώμων για το άρθρο 14 τώρα, για τις υποχρεωτικές ενδείξεις ε, και πώς θα απεικονίζονται. Πρώτα απ' όλα για την αναγνωσιμότητα των ενδείξεων. Όσον αφορά την αναγνωσιμότητα συμφωνούμε προφανώς όλοι επιθυμούν και θέλουν να είναι εύκολα εύληπτες και αναγνώσιμες οι ενδείξεις αυτές. Εκείνοι που θέλουν διαφορετικά μεγέθη γραφής ή ψηφίων να καθορίσουν πρέπει να πω σε αυτούς ότι αυτό δεν το θεωρώ ιδιαίτερα σκόπιμο και λογικό να καθορίσουμε συγκεκριμένο μέγεθος ψηφίων, διότι η αναγνωσιμότητα δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από το μέγεθος των ψηφίων. Μπορεί να έχει τρία χιλιοστά ή ενάμιση χιλιοστό ή πέντε χιλιοστά να πούμε και να είναι παρόλα αυτά μη αναγνώσιμα όταν έχουμε με ένα επίπεδο απεικόνησης ε, το οποίο στην ε, χρωματική αντίθεση ή στην αντίθεση των ψηφίων και του, της απεικόνησης των υπόλοιπων στοιχείων δεν είναι αναγνώσιμα. Ε, τα αναφερόμενα στοιχεία. Πρέπει λοιπόν αυτό σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους αλλά και σε σχέση με τις ε, οργανώσεις για την προστασία των καταναλωτών και την, ε, να είναι δια, αναγνώσιμες, εύκολα εύληπτες αυτές οι ενδείξεις. Για το άρθρο εξαιρέσεις ελάχιστων συσκευασιών σε σχέση με την υποχρεωτική ετικετοποίηση. Θα πρέπει να διεξαχθεί συζήτηση για τετραγωνικά εκατοστά αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε για το μέγεθος της, ε, της συσκευασίας πόσοι, ποιες διαστάσεις πρέπει να έχει, ώστε να δούμε πώς μπορούν όλα αυτά να καλυφθούν. Για το άρθρο 17, μη συσκευαστέντα τρόφιμα, ετικετοποίηση μη συσκευαστέντων τροφίμων. Και εδώ έχουμε διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν από πλευράς τροπολογίων, όμως υπάρχει ομοθυμία, για παράδειγμα, για την ιδέα ότι οι πληροφορίες για τα αλλογενή ή αλλεργιογόνα πρέπει να είναι διαθέσιμα, διαθέσιμες με κάποιο τρόπο σε αυτές τις συσκευασίε. Θα υπάρξει όμως αντιπαράθεση σε σχέση με την αρμοδιότητα των κρατών μελών για αυτό το σημείο. Μπορούν τα κράτη-μέλη λέει, να καθορίζουν πώς θα αντιμετωπίζονται τα μη συσκευαστέντα τρόφιμα όσον αφορά την ετικετοποίηση. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτός ο κανονισμός, αυτή η διάταξη στον νέο κανονισμό δεν θα έπρεπε να ε, εντάσσεται, να προβλέπεται. Είναι ένας ευρωπαϊκός κανονισμός και για την ενιαία εσωτερική αγορά είναι σημαντικό σε όλα τα κράτη-μέλη να έχουμε ένα ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης, πώς δηλαδή και τα μη συσκευαστέντα τρόφιμα θα αντιμετωπίζονται. Γι' αυτό είμαι κατά μια αρμοδιότητα των κρατών μελών πρωτογενώς στο σημείο μη συσκευαστέντων τροφίμων να μην είναι δηλαδή αρμόδια τα κράτη-μέλη για αυτό το θέμα στην ετικετοποίηση. Πρέπει εδώ να βρούμε μια σωστή λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πιστεύω. Τώρα, αν εξαιρέσουμε το ενόπνευμα, θα το εξαιρέσουμε ή όχι, η ενόπνευματούχα, προτείνει <clears throat> με εξαίρεση των μεικτών, των μειγμάτων αλκοολούχων ποτών να εξαιρείται το αλκοόλ, το ενόπνευμα. Θεωρώ ότι είναι θέμα του κατά πόσον θα υπάρχει μεγάλο ποσοστό αλκοόλ ή όχι, είναι αυστηρότερη ας το πούμε έτσι αυτή η ε, διάταξη. Μπορούμε ίσως ε, να συμφωνήσουμε νομίζω και σε αυτό το σημείο. Για μένα θα ήταν μια, συνεπι... μια ας το πω, συνεφαρμογή της, συνεπής, ε, ένα συνεπές συμπέρασμα αυτό για το αλκοπόψ. Υπάρχουν κάποιες ιδέες, απλά να έχουμε κάποιες εξαιρέσεις ή ειδικέ ε, περιπτώσεις για το κρασί, για τον ίνο. Αλλά υπάρχει και κάποια σκέψη το ενόπνευμα να συμπεριλαμβάνεται με αναφορά ένδειξης ε, κατόγκων. Υπάρχει και ιδέα το ενόπνευμα να αποκλείεται, να εξαιρείται αλλά να υπάρχει αναφορά ενεργειακής ε, θερμιδικής ε, ας το πω έτσι ποσότητας ε, και υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που υποστηρίζουν την έκθεσή μου ως προς αυτό και θέλουν να πούν εντάξει σωστό αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πέντε χρόνια να επανεξεταστεί η κατάσταση όπως θα έχει διαμορφωθεί αλλά μόλις ξεκινήσαμε και έχουμε μια νέα ρύθμιση για το κρασί και κατά τα άλλα πρέπει να πούμε ότι τα υνοπνευματούχα ποτά είναι, ε, δεν είναι τρόφιμα, αλλά είναι ε, ειδική κατηγορία που δεν πρέπει να ενταχθεί. Αλλά για τα αλκοπόψη μπορούμε να συζητήσουμε ούτως ή άλλως. Υποχρεωτικές τώρα αναφορές και ενδείξεις για την ε, τροφική αξία. Ποιες τροφικές ενδείξεις θα αναφέρονται. Ποιες ουσίες θέλουμε ρητά και κατηγορηματικά να αναφέρονται. Λύπη και κορεσμένα ε, λύπη, άλατα. Υπάρχουν πολλές ε, προτάσεις εδώ, πολλές ιδέες. Το θέμα είναι για το αλάτι θα αναφέρουμε το ποσοστό σε νάτριο ή θα πούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το αλάτι, το άλας να αναφέρεται ξεχωριστά. Εγώ παραμένω στη δική μου άποψη ότι το νάτριο ουσιαστικά πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά και ενδεχόμενα ως υποσημείο να έχουμε από αυτό και την αναφορά ίσως και του αλατιού διότι το αλάτι δεν είναι ακριβώς καθαρό νάτριο και έχουμε και διάφορες άλλες πηγές νατρίου στα τρόφιμα και αυτό το θεωρώ το πιο σημαντικό επιστημονικά στοιχείο αναφοράς το νάτριο. Τώρα για τεχνητά ε, προϊόντα που παράγονται θα ήθελα να πω ότι ε, τεχνητά κορεσμένα λύπη στο ε, εργαστήριο δεν είναι εύκολο να ε, διαχωρίζονται. Πώς θα το κάνουμε αυτό σε σχέση με την ετικετοποίηση των τεχνητών αυτών ουσιών λύπους. τώρα για τα ηχνοστοιχεία γιατί να μην αναφέρει αυτό έστω θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους ε, να προβληματιστούν πόσες θα είναι οι ενδείξεις. Αν έχουμε 100 διαφορετικά στοιχεία ή 100 διαφορετικές ετικέτες δεν θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Το θέμα της συνολικής απεικόνησης και έχουμε εδώ ένα σημείο με ένα χαρτάκι από μια λομπιίστρια του FDA της Βρετανικής Αρχής ε, Food ε, Foods Agency είναι αξιοπερίεργο ότι έχει διανεμηθεί κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει και τέτοιου είδους lobbying να γίνεται στη δική μας συνεδρίαση. Θα έχουμε μια χρωματική απεικόνηση όπως στους σηματοδότες της κυκλοφορίας, στους φωτεινούς σηματοδότες. Υπάρχουν λίγοι συνάδελφοι που είναι υπέρ. Εγώ πιστεύω δεν πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Θέλω σαν συνέπεια τούτου να πω ότι Πάντα εδώ πρέπει να δούμε ότι έχουμε υποχρεωτική απεικόνηση, θέμα υποχρεωτικής να σας πω γιατί είμαι εναντίον αυτών των δύο συστημάτων ή και ενός υβριδικού συστήματος, δηλαδή ενός μείγματος αυτών των δύο χρωματικών απεικονίσεων. Πιστεύω δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μπορείτε λίγη ησυχία να κάνετε συνάδελφε εσείς, παρακαλώ. Ενοχλεί πολύ να συζητάτε. Εντάξει, ευχαριστώ. Πρόεδρος, πραγματικά έχουμε μέχρι τις 11 χρόνο και ναι, με αυτό το σημείο ολοκληρώνω πρόεδρε, λέει η ομιλήτρια. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Μια χρωματική απεικόνηση ή το GDA Guided Daily Allowance ή ανάμεικτό ε, σύστημα μεταξύ των δύο. Και τα δύο συστήματα υπάρχουν σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να πω ότι από τον τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 80% όλων αυτών των επιχειρήσεων στα τρόφιμα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η μεγάλη παραγωγή, οι βιομηχανίες δηλαδή, οι μεγάλες βιομηχανίες, το GDA έχουν εισαγάγει, Guided Daily Allowance. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί την πρόταση της βιομηχανίας και προτείνει αυτό το σημείο της GDA να είναι υποχρετικό. Τώρα, εγώ είμαι κατά του να είναι υποχρεωτική αυτή η απεικόνηση, γιατί δεν έχουμε κάποιε ενδείξει πόσο ο καταναλωτή θα βοηθηθεί με αυτόν τον τρόπο πανευρωπαϊκά. Και δεν βοηθούν οι ενδείξει από ένα μικρότερο κράτο μέλο. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα όλων μα, να έχουμε ένα σύστημα απεικόνηση με το οποίο όλοι οι καταναλωτέ στα 27 κράτη-μέλη θα βοηθηθούν. Θεωρώ το σύστημα GDA ως υπερβολικά φορτωμένο. Υπερβολικά στοιχεία αναφέρονται. Είναι πολύ δύσκολα αναγνώσιμο και δεν είναι εύληπτο δεν είναι ε, χρήσιμο για την καθημερινή ζωή. Δεν μπορεί κανείς με όλη τη μέρα να κυκλοφορεί με έναν υπολογιστή και να κάνει υπολογισμούς ποια ποσοστά έχω από αυτή την ουσία ή την άλλη και ε, τι έχει γίνει σε σχέση με τα διάφορα τρόφιμα όσον αφορά αυτές τις ουσίες και τα ποσοστά τους. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα παιδιά πρέπει να λάβουμε υπόψη. Λοιπόν, είναι γνωστή η άποψή σας ήδη, μας την έχετε καταστήσει σαφή, λέει ο Πρόεδρος. Σας έδωσα επαρκή χρόνο. Έχουμε μέχρι τις 11 μόνο χρόνο οι συνάδελφοι πρέπει και τις, παρο... τις τροπολογίες τους να μπορέσουν να παρουσιάσουν. Λυπούμε Πρόεδρε, αλλά αυτό αναφέρεται στο φάκελο το σύστημα απεικόνησης με τον φωτεινό σηματοδότη, με τους φωτεινούς σηματοδότης, σηματοδότες δεν είναι λειτουργικό. Είναι παραπλανητικό και μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε πρόβλημα λοιπόν προβληματική σύντησης ε, των, ε, από πλευρά ε, των πολιτών μας αν χρησιμοποιηθεί κάτι τέτοιο. Είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα και γι' αυτό θα ήθελα λοιπόν να πω ότι έδωσα στην εισηγήτρια αυτό το χρόνο να μπορέσει να τοποθετηθεί. Θα έρθει και η Ισπανίδα υπουργό, οι συντονιστέ θα έχουν τρία λεπτά, όλοι οι άλλοι δύο λεπτά. Μετά κλείνει ο πίνακα αγοριτών και ολοκληρώνουμε. Και έτσι ούτω ή άλλω είναι στενό ο χρόνο. Βίρμοντ στην συνέχεια. Τα τρία λεπτά παρακαλώ όριο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Τη συζήτηση αυτή την έχουμε κάνει πολλέ φορέ. Θα μιλήσω για πολύ λίγα θέματα. Καταρχήν για το ενόπνευμα. Τα ενοπνευματόδη θα πρέπει να επισημένονται με τα συστατικά και τι θερμίδε, διότι δίνουν υψηλή ενεργειακή αξία στου καταναλωτέ και οι καταναλωτέ δεν γνωρίζουν την υψηλή ενεργειακή αξία των ενόπνευματοδών. Επίση, είναι σημαντικό να υπάρχει υποχρεωτική ονομασία προέλευση και για τα γεωργικά προϊόντα και για το κρέα και τα πουλιαρικά στο επεξεργασμένο, στα επεξεργασμένα τρόφιμα, γιατί είναι πληροφορίε που τι θέλουν οι καταναλωτέ και πρέπει να του τις δώσουμε. Επίση, είμαι υπέρ τη υποχρεωτική πληροφόρηση πάνω στη συσκευασία για να μπορέσει η πληροφορία να παρουσιάζεται ε, με τρόπο που θα κατανοούν εύκολα οι καταναλωτέ. Και θέλω να σα πω ότι αυτό το έντυπο το οποίο μοιράστηκε, εγώ το μοίρασα, δεν το μοίρασε κάποια ομάδα πίεση κάποιο λόμπι, όπως ε, πολύ κακώς είπε η συγγήτρια. Και είναι μια μελέτη από την υπηρεσία ε, προτύπων τροφίμων, αλλά εγώ το μοίρασα στους συναδέλφους και κανείς άλλος από ομάδα ε, λόμπι. Είναι το αποτέλεσμα μιας μελέτης 18 μηνών στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τα συστατικά των τροφίμων. Είναι η πιο συνεκτική και πλήρης μελέτη για καταναλωτικές συνήθειες σχετικά με την επισήμανση στη συσκευασία και είναι ανεξάρτητη μελέτη που έχει αξιολογηθεί από ομοτήμους. Τα αποτελέσματα λένε ότι οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν τις ετικέτες ε, τη σήμανση πάνω στη συσκευασία ε, θεωρούν ότι είναι πολύ χρήσιμες. Τις χρησιμοποιούν ιδιαίτερα αν ψωνίζουν για παιδιά και συγκρίνουν διάφορα προϊόντα ή όταν έχουν κάποια ιδιαίτερη ανησυχία για θέματα υγείας, υψηλή αρτηριακή πίεση ή διαβήτη παραδείγματος χάρη θέλουν να προσέξουν το βάρος τους. Και ε, αν υπάρχει μια τέτοια επισήμανση συνεπής, δηλαδή να υπάρχει επισήμανση στην συσκευασία, θα μπορούν να παρακολουθούν τα στοιχεία οι καταναλωτές. Ε, χρειάζεται μια ε, ετικέτα ε, που θα συνδυάζει το σύστημα του φωτεινού, χρηματο... του φωτεινού σηματοδότη και θα ε, συμπεριλαμβάνει και ποσοστά της ημερήσιας συνιστόμενης ποσότητας του GDA μαζί με τα επίπεδα θρεπτικών ουσιών σε, σε κάθε μερίδα προϊόντος. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν λέμε στους καταναλωτές τι πρέπει και τι δεν πρέπει να τρώνε. Οι καταναλωτές θέλουν τις πληροφορίες αυτές για να ενημερώνονται και δεν πρέπει να τους αρνηθούμε εμείς το δικαίωμα επιλογής. Τους καθοδηγούμε, τους δίνουμε επεξηγήσεις με τρόπο κατανοητό για να μπορέσουν να επιλέξουν πιο υγιεινές επιλογές εάν το, ε, αν το επιλέξουν. Αλλά μόνοι τους θα αποφασίσουν το τυρί και η σοκολάτα μπορεί να επισημαθούν με κόκκινο χρώμα και θα το δουν οι καταναλωτές, θα έχουν καλύτερα επίγνωση του τι καταναλώνουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Γκλένις. Κύριε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Ζόμερ, την εισηγήτρια. Σα ευχαριστούμε για τα σχόλιά σα για τι διάφορε τροπολογίες και χαίρομαι που φαίνεται ότι μερικές από αυτές μπορεί να τις δεχτεί. Και εγώ και οι συνάδελφοι προσπαθήσαμε να είμαι δημιουργική. πρέπει να δίνουμε πληροφόρηση στους καταναλωτές και όχι προ, προειδοποιητικές ε, επισημάνσεις. Αυτό είναι σημαντικό νομίζω στην τακτική που θα ακολουθήσουμε και δεν θα πρέπει να κάνουμε ένα σύστημα υπερβολικά πολύπλοκο. Όσο πιο απλό, τόσο καλύτερα. Θα πρέπει να είναι απλούστερο για τους καταναλωτές και για τους παραγωγούς. Και είναι σημαντικό να υπάρχει συνδυασμός αυτών των δύο. Πολλά σημεία θα ήθελα να συζητήσω. Και θα ξεκινήσω με αυτό το σύστημα του φωτεινού σηματοδότη στην επισήμανση. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να ενημερώνουμε του καταναλωτέ και όχι να του προειδοποιούμε και να του φοβίζουμε. Άκουσα πολύ προσεκτικά την κυρία Βίλμοντ, αλλά δεν είμαι πεπισμένο ότι το κόκκινο, το κόκκινο χρώμα για τον καταναλωτή θα σημαίνει stop τα τρόφιμα τα οποία θα έχουν κόκκινο χρώμα δεν είναι αναγκαστικά κακά για την υγεία του καταναλωτή. Η ποσότητα κατανάλωσης αυτών των τροφίμων θα είναι αρνητική ενδεχομένω. Και όσον αφορά το GDA, την ημερήσια συνιστόμενη ποσότητα, διαφωνώ με την εισηγήτρια, είναι κάτι που είναι χρήσιμο για τους καταναλωτέ. Ίσως οι επιστημονικές ε, ενδείξεις δεν είναι πάντοτε 100% σαφείς, αλλά ε, δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα στον καταναλωτή ε, η συνιστόμενη ημερήσια ποσότητα όσον αφορά τις διατροφικές τους συνήθειες. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις catering, νομίζω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε το να καταλήξουμε στο να βάζουν ανακοινώσει στα εστιατόρια και επιχειρήσεις catering που θα λέει ότι αποποιούνται πα ε, ευθύνη ε, για τα τρόφιμα τα οποία καταναλώνονται. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν την ευθύνη να ρωτάνε στα εστιατόρια τι περιλαμβάνει το μενού, οπότε θα πρέπει ο επιχειρηματίας να δίνει αυτές τις πληροφορίες όταν ο καταναλωτής τη ζητήσει. Τέλος, για τα μη συσκευασμένα τρόφιμα, συμφωνώ με την εισηγήτρια. Και τέλος, ε, για το άλλας, διαφωνώ με την εισηγήτρια. Νομίζω ότι το νάτριο δεν είναι σαφές για τον καταναλωτή, το αλάτι είναι σαφέστερο. Uh, Κύριο Σλίτερ, ευχαριστώ. Καταρχάς θα σταθώ στις ερωτήσεις της εισηγήτριας. Νομίζω για το γάλα είναι θέμα γούστου. Υπάρχει φρέσκο, ε, παστεριωμένο μα, ε, μακράς κατανάλωσης. Επομένως, ο ε, καταναλωτής έχει δικαίωμα να επιλέξει. Γι' αυτό και κατέθεσε και τη σχετική τροπολογία. Υπάρχει και η τροπολογία μου για τα παιδιά. Όλα είναι από τη Συμβάση των Ηνωμένων Εθνών. Ε, μπορεί όχι από τη χώρα σου, Ντάκμαρ, αλλά έρχονται από διάφορες από τις χώρες κάποιου. Κάποιοι πιστεύουν ότι υπάρχει. Εγώ γέλασα λίγο όταν άκουσα την ιδέα, αλλά όταν ε, μου την εξήγησαν νομίζω ότι μπορούσε να έχει κάποια αποτελέσματα. Διότι αν σκεφτείτε την οικονομία αγορά, η οικονομία αγορά βασίζεται στο γεγονό ότι έχετε τι κατάλληλε πληροφορίε για να κάνετε τι αγορέ σα. Κάποιοι είναι κατά τη παιδική εργασία, κάποιοι είναι κατά ε, ε, της των ε, αρχών εργασία. Ε, μπορεί η Κομισιόν να κάνει πρόταση και να την απορρίψουμε αν δεν ε, λειτουργεί. Αλλά γιατί να μην τους δώσουμε και τη δυνατότητα να ασκήσουν τα καθήκοντά τους και να μας παρουσιάσουν μια πρόταση. Και κατόπιν συζητάμε πάντα τη χώρα προέλευση, την προέλευση ε, των βασικών συστατικών και ούτω καθεξής. Κάποιοι λένε ότι εγώ αγοράζω από όλο τον κόσμο, δεν έχω ιδέα από πού προέρχονται και δεν έχω και καμία διάθεση να το γράφει αυτό στην επισήμαση. Ο συμβιβασμό θα μπορούσε να είναι μια, μια ε, επιχείρηση που δεν μπορεί να εντοπίσει την βασική του προέλευση να λέει αγνώστου προελεύσεω. Αυτό είναι ένα συμβιβασμό που θα μπορούσα να τον δεχτώ. Και μετά η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει. Αλλά το να λέμε απλώς ότι για κάποιους δεν υπάρχει δυνατότητα και μετά ε, θα απορρίπτουμε και τη δυνατότητα για κάποιους που γνωρίζουν από πού έρχονται τα προϊόντα τους, ε, νομίζω ότι δεν είναι υπέρ των καταναλωτών. Ε, αρμόζει στους ανθρώπους που δεν είναι και τόσο υπεύθυνοι. Ε, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να γνωρίζουν από πού προέρχονται αυτά που τρώνε το αγνώστου προελεύσεως, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι ένας κάποιος συμβιβασμός. Και μετά, κάποιες μικροαλλαγές. 3,62 για τα αυγά. Ξέρετε ότι έγινε μακρά συζήτηση και υπάρχει και το στοιχείο που μας δείχνει πώς ακριβώς, από πού ακριβώς προέρχονται τα αυγά. Ανεβιολογικά ή ούτω καθεξής. Και έχω και κάποιες τροπολογίες για το συνδετικό ιστό στο κρέας και το δεξί. Ε, παραδείγματος χάρη, οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να ξέρουν αν το 25% του κρέατος που καταναλώνουν περιέχει συνδετικό ιστό. Ε, σας παρακαλώ, εξετάστε τις τροπολογίες μου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στίβενσον θα ήθελα να συμφωνήσω απολύτως με το θέμα του εινοπνεύματος. Κυρίως την ανάγκη να υπάρχει μια κάποια συνέπεια για τον αποκλεισμό των αλκοόλουχων ποτών από αυτούς τους κανόνες. Όπως είπαμε, έχουμε ήδη κάποιους κανόνες για τον ίνο που μόλις εισήχθησαν και θα δημιουργηθεί σύγχυση στους ε, καταναλωτές αν αρχίσουμε να συμπεριλαμβάνουμε και τα υπόλοιπα ενοπνευματόδητα εδώ στους κανόνες. Πιστεύω ότι η προέκταση των κανόνων για να έχουμε επισήμανση για την περιεκτικότητα σε σάκχαρα και ενόπνευμα θα δημιουργήσει τεράστια σύγχυση. Πρέπει να γνωρίζουμε και τι θέλουν οι καταναλωτές, όπως είπε και η συνάδελφος. Οι καταναλωτές θέλουν σαφήνεια. Και αν αρχίσετε να τους λέτε, συγγνώμη Γκλέντ, αλλά εδώ θα διαφωνήσω μαζί τους. Αν αρχίσουν να τους λες πόσες ε, θερμίδε περιλαμβάνονται στο αλκοόλ, Δηλαδή, αν έχουμε την περιοπτικότητα σε θερμίδε ενό μπουκαλιού ουίσκι που εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, όταν κάνει κάποιο το συσχετισμό με ένα ποτήρι έχουμε διάφορε μετρήσεις, έχουμε ε, ε, διαφορετικές αλλαγές. Αν προσθέσουμε νερό ξέρουμε τι κάνουμε. Αν βάλετε κοκακόλα θα έπρεπε λογικά να, να μην το αποδέχεστε αυτό, να σας σοκάρει. Αλλά αυτό δεν το θέλουν οι καταναλωτές σε καμία περίπτωση. Συμφωνώ απολύτω λοιπόν με την εισηγήτρια. Ε, για λόγους συνέπειε θα πρέπει τα αλκοολούχα ποτά να μείνουν εκτό του συγκεκριμένου ε, κειμένου. Δεν είναι τρόφιμο το ουίσκι, είναι φάρμακο. Για πάσα νόσον. Επομένω, εξαιρείται από αυτήν την οδηγία. Η κυρία Λεωτάχ. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Και εμένα πραγματικά με εξέπληξε ο τεράστιος αριθμός των τροπολογιών που παρουσιάστηκαν. Θα είναι τεράστιο άχθος να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα ευανάγνωστο κείμενο για τους καταναλωτές με όλες αυτές τι τροπολογίες. Πρέπει να πω ότι είναι πάμπολε οι τροπολογίες, αλλά μεταξύ αυτών, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον κάποια σημεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο συμβιβασμό. Το πρώτο συμβιβασμό που θα μπορούσα να δεχτώ, και αυτή ήταν και ερώτηση της εισηγήτριας, αφορά την αρχή της χώρας προέλευσης. Τι εννοούσα εγώ με την τροπολογία. Συμφωνώ με τον Καρλ. Εάν δεν ξέρουμε τη χώρα προέλευση, α γράψουμε αγνώστου προελεύσεω. Εάν το γνωρίζουμε, α τη γράψουμε. Με την τροπολογία μου, αυτό που ήθελα απλώ να πω είναι ότι όπω και να έχει, ακόμα και για απλά προϊόντα, όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, γάλα, κρέα, ακόμα και για τα πιο απλά προϊόντα, κατά την άποψή μου θα έπρεπε να αναγράφεται κάπου και η προέλευση. Και για τα λοιπά προϊόντα, Α υπάρχει το βασικό συστατικό, το βασικό χαρακτηριστικό. Παραδείγματο χάρη για τη σοκολάτα περιεκτικότητα σε κακάο. Αυτό ήθελα να πω με την τροπολογία μου. Ε, εξακολουθώ παρόλα αυτά να φρονώ ότι θα πρέπει να είναι νομοθεσία υπέρ του καταναλωτή αυτή που ετοιμάζουμε. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχει κάποια προστιθέμενη αξία για τον καταναλωτή. Πολλέ οργανώσεις καταναλωτών εξακολουθούν να μας λένε ότι οι καταναλωτές προτιμούν το σύστημα του φωτεινού σηματοδότη. Εγώ θα στεκόμουν εκεί. Οποιοδήποτε σύστημα και να έχουμε, θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση. Ενώ το σύστημα του φωτεινή σηματοδότη φαίνεται να είναι κάτι το οποίο αποδέχονται οι καταναλωτές, επομένως ίσως θα έπρεπε να το ευνοήσουμε. Συμφωνώ με την εισηγήτρια, ε, ως προς τον Ίνο, αυτό θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής ε, νομοθετικής πρότασης. Ευχαριστώ. Μετά τους συντονιστές περνάμε στους υπόλοιπους αγορητές. Δύο λεπτά μόνο παρακαλώ. Ξεκινάμε με την Dagmar Rothberend. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω γοργά, σύντομα να καλύψω τα θέματα. Ξεκινώ με τις τοπολογίες που είναι οι πιο σημαντικές. Πρώτον, χώρα προέλευσης. Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν από πού προέρχονται αυτά τα προϊόντα. Και αν οι παραγωγοί λένε ότι έχουν διαφορετικές συνταγές και παίρνουν τα αμύγδαλα, ας πούμε, φέτος αυτή τη χρονιά από την Νότια Αμερική και την άλλη χρονιά του χρόνου την Ιταλία, τότε μπορώ να το κατανοήσω, θα το δεχτώ. Αλλά πρέπει να αναμένουμε ότι οι διαφορετικέ αυτέ χώρε θα απαριθμούνται, θα αναφέρονται. Χώρα πρόέλευση και μετά τρει χώρε ίσως θα αναφέρονται. Δεν έχω πρόβλημα με κάτι τέτοιο. Αναμένω όμω, α το πω έτσι, να υπάρχει εφάνταστος τρόπος αντιμετώπισης, κάλυψης. Χώρα προέλευσης, απόλυτη αναγκαιότητα πιστεύω, αδύρυτη ανάγκη να αναφέρεται. Μετά, δεν καταλαβαίνω την εισηγήτρια γιατί λέει ότι τα εχνοστοιχεία δεν είναι σημαντικά για τους ε, καταναλωτές. Έχω μία τροπολογία όπου οι πρωτεΐνες ε, και τα εχνοστοιχεία πρέπει να αναφέρονται. Υπάρχουν Πάμπολοι άνθρωποι που λόγω ασθενειών ή άλλων ευαισθησιών, ε, άλλων λόγων για την υγεία τους ε, πρέπει να γνωρίζουν τι γίνεται με τεχνοστοιχεία. Και είναι μια υποχρεωτική αναφορά αυτό. Και το να μην τους την δίνουμε αυτή την πληροφορία είναι κάτι ανησυχητικό. Έχω και μετά μια τροπολογία που έχω καταθέσει, τουλάχιστον για το κρασί και την πύρα, αλλά και όλα τα άλλα ποτά να αναφέρονται οι θερμιδικές ποσότητες ε, και οι αναλογίες. Άκουσα τι είπε ο κύριο Στίβενς πολύ προσεκτικά. Κατανοώ τι λέει και για το ουίσκι, ότι είναι συναισθηματικά φορτισμένη η κατάσταση για αυτόν, για το ουίσκι. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, κάτι τέτοιο αγαπητοί συνάδελφοι. Οι πολίτες πρέπει πραγματικά να γνωρίζουν πόσες θερμίδες έχει ένα ποτήρι κρασί και ένα ποτήρι ουίσκι. Τώρα με, κρασι... νερό ή όχι αυτό δεν αλλάζει τίποτα και υπάρχει δικαίωμα για τους καταναλωτές γι' αυτό και είναι κάτι απαράδεκτο και κανένας ε, δεν θα μπορέσει να αποτρέψει εμένα ή κάποιον να πίνει κρασί ή ε, ουίσκι και Τώρα, για να μην συμπληρώνεται κάτι τέτοιο, το θεωρώ λανθασμένο. Πρέπει να υπάρχει αυτή η ένδειξη. Και μετά, τώρα, Πρέπει να έχουμε μέγεθος ε, για τις πληροφορίες που θα είναι εύληπτο στις ε, ενδείξεις, ε. καθώς επίσης και να έχουμε ρύθμιση σε σχέση με την συσκευασία. Διαφορετικά θα υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση. Ευχαριστώ Τόμας Ούλμερ, ευχαριστώ Πρόεδρε και για την κυρία Βάις Γκέρμπερ που έχει ασθενήσει τοποθετούν. Παρ' αυτά σε δύο λεπτά θα καλύψω το θέμα για τον κύριο Στίβενσον όπως είπε ο George Bernard Shaw, είναι το ουίσκι κάτι σαν ε, μπορώ να πω φως, ε, φωτίζει τη ζωή. Τώρα για το ότι τους, στους των το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες θέλουμε να τους δώσουμε που σε μερικά δευτερόλεπτα αγοράζοντας προϊόντα μπορούν να ενημερώνονται σωστά. Αυτό είναι το εγχείρημα που πρέπει να πετύχει και δεν θέλουμε μόνο να έχουμε πολλές πληροφορίες αλλά να έχουμε επαρκείς πληροφορίες να έχει μια σωστή εικόνα για το προϊόν που αγοράζει ο καταναλωτής και να έχουμε και βελτιώσεις σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ, σε σχέση με τα νητράτα, θα ήθελα να πω ότι αυτό που έχω υπόψη είναι ότι στην, προς, στην προστινή προς όψη θα πρέπει οι, οι ουσιαστικές ε, ε, ενδείξεις να αναφέρονται και να μην υπάρχει για παράδειγμα απεικόνηση παραπλανή να μην λέγεται, να μην δείχνετε ότι κάτι είναι τυρί όταν δεν είναι πραγματικό τυρί. Και για τα GDAs εκείνο που έχω υπόψη είναι ότι επιπρόσθετα μπορούν να αναφέρονται ε, στα 100 γραμμάρια ή 100 χιλιοστόλιτρα οι ε, ενδείξεις αυτές. Δεν χρειάζεται υποχρεωτικά να υπάρχει χρωματική απεικόνηση. Μαύρο-άσπρο στην εκτύπωση μπορεί να είναι, αλλά με ένα πρότυπο όπου με διαφορετικές ενδείξεις μπορούν να ενημερώνονται οι πολίτες ε, γραφικά δηλαδή, με το γράφημα αυτό, την απεικόνηση. Υπάρχουν διάφορα πρότυπα. Αντίστοιχα έχω αναφερθεί στις τροπολογίες μου σε αυτά τα πρότυπα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πέτερ Λίζε παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στις ε, πολλές εκατοντάδες τροπολογίες, μία μόνο, μόνη είναι δική μου που έχω καταθέσει εγώ. Η έκθεση θεωρώ ότι είναι μια καλή βάση. Όμως έχω μία τροπολογία και θέλω να επεξηγήσω περί τίνος πρόκειται αυτή η τροπολογία μου. Συζητήθηκε και αναφέρθηκε ότι τα μη συσκευασμένα τρόφιμα θα θέλαν κάποιοι να εξαιρεθούν, τουλάχιστον όσον αφορά τις ε, ευρύτερες υποχρεώσεις ε, ενδείξεων όχι όσον αφορά για παράδειγμα τις, ε, τα ουσιώδη συστατικά αλλά τις θερμίδες ή τα κορεσμένα λίπη ή μη κορεσμένα λίπη. Αυτό σίγουρα είναι δύσκολο για μικρές επιχειρήσεις να γίνει και θα ήθελα αυτό να το επεκτείνω, να το διευρύνω κάπως. Υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις που προσφέρουν συσκευασμένα τρόφιμα σε ένα ή δύο σημεία. Για παράδειγμα ένας γεωργός που όχι μόνο ο ίδιος ε, στην εκμετάλλευση το κάνει αυτό, αλλά δίνει και σε ένα γειτονικό ξενοδοχείο τα λουκάνικα που παράγει ο ίδιος αυτός αν αυτή την δημιουργικότητα σε σχέση με τις μικρές επιχειρήσεις ή και με τους χασάπιδες ή και με τους αρτοπιούς, αν υποχρεώσουμε όλους αυτούς τους μικροπαραγωγούς να κάνουν αυτά που έχουμε υπόψη να κάνει η Φεραίρο και η Νέσλε, οι μεγάλες επιχειρήσεις, τότε θα είναι ασφικτικά τα πλαίσια για την δημιουργικότητά τους. Στο, τα Χριστούγεννα παράγεται κάτι διαφορετικό, ειδικό προϊόν. Και αν πούμε ότι αυτά με τα κεκορεσμένα ή τα μη κεκορεσμένα και τι θερμίδε πρέπει να αναφέρονται, ε, τότε αυτή η μικροπαραγωγή θα πούν εντάξει δεν μπορώ να τα καταφέρω πια, θα τα παρατήσω και έτσι θα είναι ασφικτικό αυτό, στραγγαλιστικό για αυτούς. Μετά, τελευταία μου παρατήρηση για τη χρωματική απεικόνηση και εγώ πιστεύω ότι είναι προβληματικό να είναι υποχρεωτικό κάτι τέτοιο για πανευρωπαϊκή χρήση υπήρξε καγχασμός, καγχάσαν κάποιοι όταν είπε η Ρενάτε Ζόμερ ότι μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη διατροφή κάτι τέτοιο. Υπάρχουν όμως και άλλες καταστάσεις. Για τους ε, πρεσβύτες για παράδειγμα, τους υπερήλικες, ε, υπάρχει το πρόβλημα να παίρνουν πολύ λίγες ε, θερμίδες και το κόκκινο σημαίνει Λοιπόν, stop εδώ, υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, κάτι τέτοιο μπορεί να είναι προβληματικό για αυτούς. Ευχαριστώ. Αντώνιο Χανόβα παρακαλώ. Κυρία Παρφανόβα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατέθεσα τροπολογίες και όλα αυτά συνάδουν με τις πληροφορίες που δίνονται στους καταναλωτές και ε, κυρίως το αλάτι, η ζάχαρη και τα λιπαρά. Αυτά ενδιαφέρουν τους καταναλωτές και την υγεία τους. Όταν μιλάω για, με συναδέλφους, ε, γιατρούς και καθηγητές βιοχημίες, πραγματικά τους οι συζητήσεις που κάνουμε εμείς εδώ και λένε ότι είναι απίστευτο οι ευρωβουλευτές να μην ε, να πάρουν ε, επαγγελματική εμπειρογνωμοσύνη και θεωρούν ότι τα αλκοολούχα ποτά δεν είναι τρόφιμα και θεωρείται τρόφιμο το αλκοολούχο ποτό από τότε που η διαιτολογία ε, έγινε επίσημη επιστήμη. Η περιεκτικότητα χάρου στο αλκοόλ έχει σημασία Οτιδήποτε και να προσθέσουμε, νερό, πάγο, είναι πολύ σημαντικό ο να γνωρίζει ποια είναι η μερίσια πρόσληψη σε ζάχαρη. Επίσης, όταν μιλάμε για το φωτεινό σηματοδότη, αυτό που έχει σημασία είναι ποια είναι η μερίσια πρόσληψη και η ε, ατομική πρόσληψη άλατος. Εχθές, αν θυμάστε καλά, η υπουργό είπε ότι θα ξεκινήσει μια εκστρατεία για την μείωση της κατανάλωσης άλατος, γιατί δημιουργεί ε, καρδιακές παθήσεις, υψηλή πίεση και είναι επικίνδυνο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα κόκκινο, γιατί είναι σήμα προειδοποίησης, δεν είναι απλώς ενημερωτικό. Πρέπει να είναι σε κόκκινο για μας, γιατί σώζει ζωής. ζωές. Δεν απλώς αθώες ε, πληροφορίες. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δίνουμε στον καταναλωτή για να είναι ενήμερος για τους κινδύνους για την υγεία του. Γιατί οποιαδήποτε τρόφιμο παίρνουμε έχει σημασία γιατί αφορά στη βιοχημία του σώματός μας. Ευχαριστώ πολύ. Ποτέ δεν ε, θα θεωρείτε μόνο θέμα κακής διατροφής. Έχω δει ε, μόνο ανθρώπους που πάσχουν από συγκεκριμένη ε, ε, διαταραχή διατροφής που μπορεί να μην αγοράζουν κάποια τρόφιμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια σειρά τροπολογιών κατέθεσα. Θέλω να τονίσω ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα που πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, προβληματίστηκε επαρκώς τι πρέπει να γίνει, διότι δεν πληρώνουν πολλοί τελικοί καταναλωτές για τέτοιου είδους προϊόντα. Κάνω λόγο για παράδειγμα για ασθενείς σε νοσοκομεία συχνά συσκευασμένα γεύματα τους δίνονται. Αυτοί ακριβώς οι καταναλωτές πρέπει να έχουν το ίδιο δικαίωμα, να έχουν εύκολα προσπελάσιμες πληροφορίες όπως οι άλλοι που αγοράζουν κάτι σε ένα μαγαζί. Έχω δύο τροπολογίες που κατέθεσα, 286-289 προσπαθούν ακριβώς τουλάχιστον αυτή την ομάδα καταναλωτών να την ενδυναμώσουν στο δικαίωμά τους, να παίρνουν αυτές τις πληροφορίες, να την ενισχύσουν. Διότι για τους παραγωγούς δεν υπάρχουν μεγάλα εμπόδια ή δαπάνες αυτά τα προϊόντα να ετικετοποιούνται όπως πρέπει όπως ακριβώς και τα άλλα που αγοράζονται σε υπεραγορές, σε σούπερ μάρκετ, ώστε οι υπερήλικες και οι ασθενείς να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους έτσι. Θέλω αυτό λοιπόν να καλυφθεί έτσι, επειδή κανείς άλλος δεν ε, αναφέρθηκε σε αυτό. Εργάστηκα πολύ στο παρελθόν σε σχέση με τρόφιμα και όσον αφορά και τα θέματα καταναλωτών και πολιτών όσον αφορά τα τρόφιμα. Ένα θέμα το οποίο συχνά διαρκώς αναφέρεται ότι πρέπει να είναι εύληπτες οι πληροφορίες και εύκολα αναγνώσιμες ε, οι πληροφορίες στη συσκευασία. Και για όσα αναφέρονται και λέγονται. Πρέπει να ξέρει κανείς αν έχει ε, διακορε... υπερκορεσμένα λύπη ένα προϊόν ή όχι. Και θέλουμε να έχουμε στην ετικετοποίηση σχετική αναφορά. Τώρα, όσον αφορά τη συζήτηση για το αλκοόλ, για το, το, τα εινοπνευματόδη, με εκπλήσει κάπως ε, η Σουηδία θέλει να έχει πιο αυστηρές διατάξεις ε, για το ενόπνευμα, διότι υπάρχει εθισμός σε σχέση με την κατανάλωση ενόπνευμα Εντάξει, αν συμβαίνει λοιπόν κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να εντάσσεται αυτό στις διατάξεις που εδώ τώρα εγκρίνονται. Πράγμα το οποίο ισχύει για τα γενικά, τρόφιμα, γενικά για τα τρόφιμα. Δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικά μηνύματα για τέτοια. Η συγγήτρια κατέθεσε μια πολύ καλή πρόταση και σε πολλά πράγματα μπορώ να συμφωνήσω μαζί της. Ένα πράγμα όμως δεν πρέπει να κάνουμε πιστεύω. Εδώ η πρόταση εθνικές ρυθμίσεις ε, ότι μπορούν να εισαχθούν. Είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Αυτό πάλι διακυβεύει την ενιαία εσωτερική αγορά. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε οι κανόνε, οι διατάξει αυτέ να είναι πανευρωπαϊκέ, πανευρωπαϊκού χαρακτήρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, για την ένδειξη χώρα προέλευση, κυρίε και κύριοι, για το κρέα ή για τα επιμέρου προϊόντα, μπορώ να φανταστώ πολύ καλά ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και το ρυθμίζουμε έτσι. Τι να αναφέρουμε όμω με πολλέ χώρε σε σχέση με ένα προϊόν που έχει 20-30 συστατικέ ουσίε να αναφέρουμε μεταφέρουμε όλες τις χώρες προέλευσης αυτών. Σε τι ωφελεί για την ενημέρωση πληροφοριών να πούμε, των πολιτών. Να πούμε ε, Κολομβία για το ένα, Μπουρκίνα Φάσο για το άλλο. Αυτά δεν ενδιαφέρουν τους ε, πολίτες ούτως ή άλλως, τους καταναλωτές. Δεν πρέπει την αλυσίδα αυτή πληροφοριών να την υπερβαρύνουμε πολύ. Έχω διαφορετική άποψη λοιπόν από την κυρία Ροτ Μπέρεντ. Για τα, ενο, για τα το, ε, εδώ είναι, αποκλίνουν οι απόψεις. οι Πρέπει να ρυθμίσουμε το θέμα των υνοπνευματοδών, έχουμε όμως και χωριστές διατάξεις για το κρασί και είναι σημαντικό να το λάβουμε αυτό υπόψη. Εδώ λοιπόν να σκεφτούμε μήπως ε, θα θέλαμε να εντάξουμε αυτά τα προϊόντα σε ετικετοποίηση. Θέλω να κρούσω κόδωνα κινδύνου όμως και συμφωνώ με τον κύριο Λίζε ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για την εισαγωγή τέτοιων κανόνων και διατάξεων ως υποχρέωση για τους μικρούς παραγωγούς και τώρα να πούμε σε όλους αυτούς τι ακριβώς πρέπει να επισημαίνουν. Αυτό θα υπερβαρύνει γραφειοκρατικά ε, τις επιχειρήσεις που έχουν 5 ή 10 για το πολύ πολύ ε, εργαζομένους που ούτως ή άλλως πρέπει να τηρήσουν κάποιες διατάξεις και υποχρεωτικού χαρακτήρα. Να υπερβαρύνουμε λοιπόν αυτά τα πλαίσια δεν είναι καθόλου θετικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κορίν Λεπάζ. Euh, Συμφωνώ με την τροπολογία της κυρίας Βίλμοντ. Αλλά θέλω να θέσουμε το πρόβλημα ξεκάθαρα. Δηλαδή, τι θέλουμε, ποιο είναι ο στόχο αυτή τη νομοθεσία. Αυτό που θέλουμε, και το υπενθύμησε και η κυρία Ροτ Μπέρεντ προηγουμένω, είναι να μπορούν οι Ευρωπαίοι καταναλωτέ να γνωρίζουν περί τίνο πρόκειται, να γνωρίζουν και τα προβλήματα υγεία που έχουν και με βάση ε, τον τρόπο ζωή του να μπορούν να επιλέξουν τα τρόφιμα τα οποία θα καταναλώνουν. Άρα, εμεί πρέπει να του δώσουμε μία επισήμανση που θα του δίνει τη δυνατότητα να κάνουν ακριβώ αυτό. Και δεν νομίζω ότι πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από φόρου, ότι ο κακομοίρη, ο καταναλωτή αισθάνεται υποχρεωμένο να κάνει κάτι ή ο κακομοίρη, ο καταναλωτή φοβάται για να υπεραμεινθούμε τελικά συμφερόντων που δεν είναι καθόλου τα συμφέροντα των καταναλωτών πρέπει να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αν η κατεύθυνση αυτή είναι αυτό το οποίο λέμε ότι κάνουμε, δηλαδή το συμφέρον του καταναλωτού, αυτό θα πρέπει να επιτρέπει και η επισήμανση. Είτε όσον αφορά ε, τις επιπτώσεις του άλατος, του, της ζάχαρης ή των ε, θερμίδων, της ενεργειακής αξίας, είτε όσον αφορά το θέμα της ονομασίας προέλευσης αν θέλουμε να κρατήσουμε μια σχέση μεταξύ της προέλευση των προϊόντων ώστε να είναι προϊόντα που προέρχονται από την ε, κοντινή περιοχή, θα πρέπει να δίνουμε στον καταναλωτή τη δυνατότητα να το επιλέγει. Αλλιώ συμφωνώ με τον κύριο Σλίτερα. Άμα δεν ξέρουμε από πού έρχεται, λέμε αγνώστου προελεύσεω. Αν δεν ξέρουμε, να, να το δηλώνουμε. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε εμείς και να κάνουμε αυτό το οποίο όντω θα επιλέξουμε. Να μην επιλέγουμε προφάσει για να κρύψουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, αν είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο δηλώνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω από την ε, Προεδρία να συζητήσουμε ξανά το θέμα σε άλλη μια συνεδρίαση, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Όσον αφορά στην επισήμανση, συμφωνώ πολύ με την εισηγήτρια. Δεν μπορούμε να βάζουμε τεράστιου χαρακτήρες σε ένα σοκολατάκι ή σε ένα πακέτο μακαρόνια. Είναι προφανές ότι είναι περιορισμένο ο χώρος που μπορούμε να γράψουμε. Υπάρχουν προβλήματα και για τους, ε, τους τροφίμων αλλά και για τους καταναλωτές. Να ρωτήσω το εξή. γιατί εγώ δεν πρέπει να ξέρω αν τα μήλα που αγοράζω προέρχονται από την Αργεντινή που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα ή παρασιτοχτώνα διαφορετικά από αυτά που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη και γιατί να μην μπορώ να επιλέξω ένα ιταλικό μήλο εάν δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος να αναγράφει επάνω αν είναι από την Αργεντινή, από την Ιταλία ή από την Ευρώπη εν γέννη. Είναι δικαίωμά μου να διαλέγω για το γιο μου το μήλο που θέλω. Υπότιτλοι AUTHORWAVE ή θα υπάρχει συγκεκριμένο κανόνες όπου συγκεκριμένες ουσίες ε, επικίνδυνες για μας θα απαγορεύονται ή θα πρέπει να έχω δικαίωμα να επιλέξω το ένα προϊόν αντί του άλλου. Όσον αφορά στο φωτεινό σηματοδότη, συμφωνώ απολύτως με την ε, εισηγήτρια. Θεωρώ ότι είναι επικίνδυνος ο φωτεινός σηματοδότης. Σκεφτείτε ένα προϊόν που περιλαμβάνει ζάχαρη ή ε, κάποια χρωστική ουσία. Θα μπορούσε κάποιο να το επιλέξει αντί κάποιου άλλου. Παραδείγματο χάρη, ένα προϊόν με ζάχαρη θα έχει κόκκινο σηματοδότη. Ενώ ένα ε, ε, προϊόν με χρωστική ουσία ε, θα είχε πράσινο, αλλά ξέρουμε όλοι ότι έχει επιβαρυντικέ συνέπειε. Παραδείγματο χάρη απαγορεύεται για τι έγκυε γυναίκε. Εμεί όμω θα βάλουμε κόκκινο και θα το απαγορεύουμε για τις για τη ζάχαρη και θα έχουμε πράσινο που απαγορεύεται για τις εγγύου ένα προϊόν με χρωστική ουσία. Σκεφτείτε για παράδειγμα τα γλυκά. Γλυκά που περιλαμβάνουν ε, χρωστικές ουσίες και σακχαρούχα προϊόντα και άλλα ε, που περιλαμβάνουν ζάχαρη. Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο αν θέλουν μπορεί να κρατήσουν τους κανόνες γιατί άλλωστε υπάρχουν κανόνες που επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να έχουν επιπλέον επισημάνσεις. Αλλά δεν μπορείτε να επιβάλλετε στην Ευρώπη τους κανόνες σας. Η Πιλάρα Γιούζου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Καταρχάς να συγχαρώ την εισηγήτρια. Εξαιρετική έκθεση που μας παρουσίασε. Συμφωνώ απολύτως μαζί της με το θέμα του φωτεινού σηματοδότη. Παραδείγματος χάρη για τον Ίνο. Το ίνο και τα, ο ίνος και τα αλκοολούχα ποτά περιλαμβάνουν τις περισσότερες νομοθετικές ρυθμίσεις για οποιοδήποτε προϊόν που χρησιμοποιούμε στην, ε, στο μπουκάλι υπάρχει και η περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Εγώ όταν λοιπόν παίρνω ένα μπουκάλι ουίσκι ξέρω πόση ποσότητα αλκοόλ λαμβάνω γιατί ε, αναφέρονται οι βαθμοί στην, ε, στο μπουκάλι. Στο θέμα της προέλευσης. Το εξήγησε και ο κύριος Σόμερ. Τα προϊόντα τα οποία ε, προέρχονται από διάφορες χώρες, περιέχουν διάφορες συστατικά από διάφορες χώρες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρουμε από πού προέρχεται το καθένα. Επίσης μπορεί να υπάρχει και θελουσία επισήμανση από τον παραγωγό, ο οποίος μπορεί να γράφει την προέλευση και έτσι να κερδίσει περισσότερα από ένα προϊόν. Και επίσης να πω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για εξαντλητικές πληροφορίες που να περιλαμβάνουν τα πάντα. Θέλουμε να ενημερώνουμε το μέσο καταναλωτή με έναν τρόπο που θα είναι καθόλου κατανοητός για αυτόν και επίσης δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε ε, με κόστος ε, τις επιχειρήσεις. Να μην ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη το μεγαλύτερο τμήμα του διατροφικού κλάδου είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντέξουν το επιπλέον κόστος που μπορούν να αντέξουν οι τρεις ή τέσσερις μεγάλες πολυεθνικές οι οποίες Ε, ε, μπορούν να αντέξουν ένα αντίστοιχο κόστος. Ε, Τίποτα επιπλέον από πλευράς μου. Να συγχαρώ για άλλη μια φορά την εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Άννα Μπίλτ τελευταία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά που με καλώς όρισατε στην Επιτροπή σας σήμερα. Είναι καλό να βλέπει κανείς ότι οι περισσότεροι από εμάς συμφωνούν πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία προστατεύοντας τον καταναλωτή, αποφεύγοντας να δημιουργήσουμε υπερβολική γραφειοκρατική υπερβάρυνση για τις, τους μικρούς παραγωγούς και να εναρμονίσουμε την ενιαία αγορά χωρίς να έχουμε προσκόμματα και εμπόδια. Εγώ θέλω λοιπόν, μια και η έκθεση αυτά τα λαμβάνει υπόψη, να υποστηρίξω αυτά τα αιτήματα. Μια και πιέζει ο χρόνος να επικεντρωθώ σε ένα θέμα. Εδώ θέλουμε να δώσουμε δώσουμε δικαιώματα στους καταναλωτές, ε, να υπάρχει η εύληπτη, ευανάγνωστη, σωστή ενημέρωση, ώστε να μπορούν ελεύθερα να επιλέγουν τα προϊόντα που επιλέγουν. Να σεβόμαστε την πολυμορφία. Εδώ θέλουμε να ενημερώνουμε, όχι να κυδεμονεύουμε και να καθοδηγούμε. Και ρωτώ την κυρία Βίλμερ, πώς μπορούμε να καθοδηγήσουμε και ταυτόχρονα να τους αφήνουμε ελεύθερους να αποφασίζουν για τον εαυτό τους τι θέλουν. Αντίφαση είναι αυτό. Εμείς οι πολιτικοί πρέπει να ενημερώνουμε, να μην επιλέγουμε τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες. Έχουν το δικαίωμα της ελευθερίας επιλογής οι πολίτες. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που πρέπει να διαφυλαχθεί αυτό και γι' αυτό οτιδήποτε ε, δίνει στους ανθρώπους μικρό επίπεδο σεβασμού, σεβασμού και αποδοχή των επιλογών τους είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Συνεχίζω να ταΐζω με βούτυρο το παιδί μου που είναι 5 ετών. Περιέχει βιταμίνη α. Φυσικά δεν θα παίρνω εγώ την ίδια ποσότητα που παίρνει το παιδί. Εμείς οι γυναίκες δεν πρέπει να υποχρεώνουμε τα παιδιά μας να έχουν ε, διαιτολόγιο με ε, χαμηλά ε, νιτράτα με μικρές ποσότητες αυτών των ουσιών. Υπάρχει μια μελέτη που έχει τυπωθεί στην Αγγλία. Δεν ανταποκρίνεται στα 500 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μόνο στο τι γίνεται σε σχέση με την Αγγλία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν αυτό το στοιχείο, να σεβόμαστε τι επιθυμούν οι πολίτε. Ευχαριστώ, Σα ευχαριστώ. Την κυρία Γκαρτίνη την, την ξεχάσαμε, έχει τον λόγο τώρα παρακαλώ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, είχα ζητήσει το λόγο, δεν με είδατε, δεν πειράζει. Ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια διότι έχει κάνει τεράστια δουλειά, αλλά θα ήθελα επίσης να πω ότι αυτό που ουσιαστικά πρέπει να συζητήσουμε εδώ είναι τι προσέγγιση θέλουμε να ακολουθήσουμε. Είναι σαφές ότι υπάρχουν ε, ρίζουσες απόψεις, είναι σαφές ότι υπάρχουν αυτοί που θέλουν να εκπαιδεύσουν τον ε, καταναλωτή και αυτοί που θέλουν απλώς να τον ενημερώνουν. Παραδείγματο χάρη, στην Ιταλία όπου ξέρετε ότι το θέμα της διατροφής είναι κάτι που είναι στο DNA μας, υπάρχουν ε, ήδη στις εφημερίδες οι τίτλοι για την προσέγγιση που θεωρείται ότι είναι λίγο παραπάνω τυπικός από όσο πρέπει και ε, μιλήσαμε ακόμα και στην επιστροφή στα, στους ηθικούς κανόνες που θα επιβάλλουν στους ανθρώπους τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν. Η προσέγγιση λοιπόν, όπως αυτοί που μας ζητούν ε, κάποιοι συνάδελφοι, είναι λίγο επικίνδυνη. Τα φωτάκια, όλα αυτά, κόκκινο, πρασινάκι, ξέρω εγώ, μπορεί να δημιουργήσει πραγματικά στρεβλώσεις. Σκεφτείτε τις ε, διατροφικές διαταραχές. Εμείς έχουμε πάμπολες κοπέλες οι οποίες ε, σπρώχνονται προς την ε, ανορεξία. Αν βάλουμε κόκκινο στο αλάτι, στη ζάχαρη, στα λιπαρά, ναι μεν ότι πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο, αλλά πρέπει να τα προσλαμβάνει το σώμα μιας έφηβης γυναίκας. Υπάρχουν έφηβες κοπέλες οι οποίες τα απορρίπτουν από την καθημερινή τους διατροφή. Ε, εμάς μας παρακολουθούν παιδίατροι από τότε που γεννιούνται τα παιδιά, που εκπαιδεύουν τις μητέρες και τα παιδιά πώς να διατρέφονται σωστά μπορούμε να διαχειριστούμε κάποιες απλές πληροφορίες που δεν θα είναι πάντα ένα σήμα κινδύνου. Οι τελευταίες έρευνες που έγιναν καταδεικνύουν ότι οι καταναλωτές ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να διαχειριστούν τη διατροφή τους ε, και είναι λίγο σαφή τα πράγματα. Μην υπερβάλλονται. Ε, τα διατροφικά προφίλ ε, κατά την άποψή μου είναι υπερβολικά και εγώ νομίζω ότι είναι σωστή η τροπολογία 162 της κυρίας Σόμερ που ξέρουμε ότι Υπάρχουν κάποια πράγματα στον 124 του 2006 για τα διατροφικά στοιχεία. Δεν θα επεκταθώ άλλο. Ε, συμφωνώ με την πρόταση του κυρίου Ρώση να κάνουμε άλλη μια συνεδρίαση γιατί είναι πάρα πολλά τα πράγματα που έχουμε να συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Πολύ καλά. Το θέμα ήδη είναι κάτι το οποίο το έχουμε, έχουμε εξοικειωθεί με αυτό για εκείνους που ήταν παρόντες την τελευταία φορά. Έχουμε το ίμιση των τροπολογιών σε σχέση με την, ε, τον αρχικό αριθμό. Μπορούμε λοιπόν να τα δούμε αυτά. Τώρα θα λάβει τον λόγο η συγγήτρια πάλι. Παρακαλώ να συγχωρέσει η Επιτροπή διότι περιμένει εκτός εθούσης η Ισπανίδα Υπουργό. Τρία-τέσσερα λεπτά το πολύ πολύ κυρία Ζόμερ για να καλύψετε κάποιες συγκεκριμένες πτυχές αν θέλετε. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω μια επισήμαση για τη μορφή απεικόνησης. Για GDA ή σύστημα σηματοδοτών ή ένα υβριδικό σύστημα μεταξύ των δύο. Αυτό που θέλω είναι να μην είναι υποχρεωτική η απεικόνηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με αυτόν τον τρόπο. Επειδή δεν ξέρουμε τι θα κάνει και τι μπορεί να κάνει ο καταναλωτής με τέτοιου είδους πληροφορίες. Όταν διαβάσετε την έκθεσή μου θα το δείτε αυτό ξεχωριστά. Τώρα, επιτρέψτε μου να επιτρέψουμε μια ε, ε, εθελοντική, εθελούσιου χαρακτήρα ε, απεικόνησης ή ένδειξης, επαναλαμβάνοντας ενδεχόμενα κάποια στοιχεία με αριθμούς ε, ή με απεικόνηση. Είναι σωστό να μπορεί να αποφασίζει τελικά ο ίδιος ο καταναλωτής ποιο σύστημα χρειάζεται, ποιο μπορεί να χρησιμοποιήσει και ποιο είναι εκείνο το οποίο θα μπορέσει να είναι θετικό. Και έτσι αυτό θα χρησιμοποιείται. Παραμένω στην την άποψή μου ότι δεν θέλω να έχουμε επιπρόσθετα εθνική, ε, ακόμα και μη δεσμευτικού χαρακτήρα, εθνική επισήμανση, ετικετοποίηση. Όπως και δεν θέλω να επιτραπεί τα κράτη-μέλη να μπορούν να αποφασίζουν το τι θα γίνει με μη συσκευασμένα τρόφιμα. Ε, αναλαμβάνω, είναι ευρωπαϊκός κανονισμός και ευρωπαϊκή ρύθμιση. Πρέπει εδώ να ρυθμίζεται και να ισχύει ενιαία στα κράτη-μέλη αυτό. Αλλά τώρα για την ε, εθελοντική επισήμανση, απεικόνηση από τον τομέα τομεακά μπορεί αυτή να επιτρέπεται. Στην κυρία Ροτ Μπέρεν να πω ότι για τις κυριότερες συστατικές ουσίες ε, ε, υπάρχει εδώ δυσκολία δυσκολία απεικόνησης ε, όμως για πρακτικούς λόγους, ε, παρότι αυτό θα ήταν ίσως ευταίο, να μπορέσουμε να αποφύγουμε να γίνεται. Μπορείτε να δείτε τι γίνεται στις ε, εταιρείε παραγωγούς ε, αυτά τα προϊόντα και θα δείτε το πώς λειτουργούν τα πράγματα. Και ταχύτατα θα αναγνωρίσετε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό να γίνει, να αναφέρονται οι κυριότερες συστατικές ουσίες, εκτός από το να επιτρέψουμε, αν επιτρέψουμε πρόσθετες ετικέτες ή επιπρόσθετα τα αυτοκόλλητα να χρησιμοποιούνται στα ε, τρόφιμα. Και υπάρχει όμως εδώ διαδεδομένη άποψη ότι πρέπει να είναι τυπωμένα αυτά πάνω στις συσκευασίες, οι υποχρεωτικές ενδείξεις δηλαδή. Και τώρα για την προέλευση των στοιχείων αυτή δεν αλλάζει αετήσια, μπορεί και αναημέρα να αλλάζει η προέλευση αυτών των συστατικών ουσιών. Και αυτό είναι ιδιαίτερα κάτι που για τον μικρομεσαίο τομέα, για τους, τις μικρές επιχειρήσεις δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθούν με τέτοιου είδους υποχρεώσεις. Σύμφωνα με τη δική μου πείρα σε σχέση με διαφορετικές τέτοιες ενδείξεις και συσκευασίες με την αλλαγή της καθημερινής προέλευσης αυτών των ουσιών είναι υπερβολική επιβάρυνση και πρέπει εδώ να δούμε και τις διαφορετικές γλώσσες ε, που πρέπει να αναφέρονται γλωσσικά πάνω στις ετικέτες. Δεν γίνονται λοιπόν όλα αυτά, δεν μπορούν να γίνουν. Δεν θέλουμε να ε, δημιουργούμε σκουπίδια από πλευράς ετικετοποίησης που θα είναι άχρηστα δηλαδή για τους καταναλωτές. Ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Μπορώ να σας διασφαλίσω ότι είμαι πράγματι πρόθυμη να συμβιβαστούμε και να συζητηθούμε. Αν θέλετε κάτι για να υπάρξει συμβιβαστική τροπολογία, να έρθετε σε μένα να το συζητήσουμε. Είμαι πρόθυμη να καταλήξω σε τροπολογίε συμβιβαστικέ για την ψηφοφορία που θα έχουμε το Μάρτιο στην Επιτροπή μα. Ευχαριστώ. Μάλιστα, σα ευχαριστώ κυρία Ζόμερ. Είναι ένα φλέγον θέμα αυτό που πάρα πολύ. Ε, έντονα έχει συζητηθεί με ε, τριβές και ε, ε, αντιπαραθέσεις όπως έχει καταστεί σαφές. Στις 16 Μαρτίου θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε αυτά τα θέματα πράγμα το οποίο, για ένα θέμα το οποίο εκκρεμεί από την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Είναι πρόθυμη διμερώς να έρθει σε επαφή με συντάκτες τροπολογιών η συγγήτρια, με την κυρία Γκαρντίνη και άλλους και άλλες, για να εξευρεθούν συμβιβαστικές τροπολογίες ή δυνατόν. Εντάξει, σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση που κάναμε. Ζητώ συγγνώμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν θα είναι δυνατόν να ακούσουμε, δεν ήταν δυνατόν να ακούσουμε τη δική της παρέμβαση και τοποθέτηση και έχουμε το τελευταίο τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη με την Ισπανίδα Υπουργό Περιβάλλοντος τώρα που πρέπει να καλύψουμε. Είχαμε πει ε, κάποια λεπτά, με κάποια λεπτά καθυστέρηση. Ε, λοιπόν, θα περιμένουμε ένα-δύο λεπτά μέχρι ότου η αντιπροσωπεία να προσέλθει στην αίθουσα. Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, αν θέλετε να καθίσετε πάλι όλοι στα έδρανά σας και ίσως να σταματήσετε να συνομιλείτε, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι με την ημερήσια διάταξη, με ένα σημαντικό σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι το πρόγραμμα της Ισπανικής Προεδρίας όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη χαρά είναι για μένα να καλωσορίσω την Προεδρεύουσα του Συμβουλίου Υπουργό Περιβάλλοντος της Ισπανικής Κυβέρνησης, την κυρία Ελένα Εσπινόσα. Κυρία Υπουργέ, καλώς ήρθατε θερμά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μία από τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές επιτροπές που έχουμε εμείς στο σώμα των εκλεγμένων αντιπροσώπων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολλούς συναδέλφους που και στις χώρες τους ε, ιδιαίτερες προσπάθειες καταβάλουν για την προσπάθεια του περιβάλλοντος πανευρωπαϊκά. Και έτσι έχουμε πάρα πολλά θέματα, πληθώρα θεμάτων που πρέπει να συζητηθούν. Καλώς ήρθατε λοιπόν θερμά. Σας δίνω αμέσως τον λόγο για την παρουσίαση του προγράμματος της Ισπανικής Προεδρίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, Έρχομαι εδώ στην Επιτροπή σας για να σας ενημερώσω για το πρόγραμμα εργασίας της Ισπανικής Προεδρίας. Παρά το γεγονός ότι είναι προφανές ότι η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και ο καθορισμός των βημάτων που πρέπει να κάνει η Ευρώπη είναι προτεραιότητα για μας αυτό το εξάμεινο, στις 20 Ιανουαρίου Εξήγησα ήδη ενώπιον του Κοινοβουλίου τα αποτελέσματα της διάσκεψης της Κοπενχάγης και τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη διάσκεψη. Δεν θα ήθελα λοιπόν εδώ να επαναλάβω τα ίδια πράγματα, αν και θα ήθελα να επισημάνω το ενδιαφέρον των 27 Υπουργών Περιβάλλοντος για την εφαρμογή άμεσα του περιεχομένου της ε, Συμφωνίας της Κοπενχάγης. Θέλουμε να προχωρήσουμε με γρήγορους ρυθμούς αποτελεσματικά για την Διεθνή Σύμβαση η οποία θα γίνει στην επόμενη διάσκεψη της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών που θα γίνει στο Μεξικό τον επόμενο Νοέμβριο. Σε κοινοτικό πλαίσιο Θέλουμε να προωθήσουμε την ενσωμάτωση μέτρων προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές σε πολύ σημαντικές πολιτικές, όπως για παράδειγμα η προστασία του εδάφους, η αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων, ε, η βιοπικιλότητα και φυσικά η γεωργία και η αλία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η Ισπανία στη διάρκεια του εξαμήνου της Προεδρίας της θα προάγει και θα προωθήσει τις εργασίες ε, της λεγόμενης Λευκής Βίβλου για θέματα προσαρμογής. Το ενεργειακό πακέτο και το πακέτο των κλιματικών αλλαγών, τα οποία το επόμενο χρονικό διάστημα θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την καταπολέμηση του φαινομένου, κυρίως στον κοινοτικό άξονα του εμπορίου δικαιωμάτων εκπομπών, θα αποτελέσει βασικό πυλώνα της πολιτικής μας. Πριν κλείσω το σημείο αυτό, θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντική σχέση έχει η εσωτερική μας πολιτική και η διεθνής ε, πολιτική και ο συνδυασμός τους. Τα μέτρα που υιοθετούμε περιλαμβάνουν την ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο θέμα αυτό, αλλά οι διεθνείς σχέσεις μπορεί να χρειαστούν και κάποιες προσαρμογές ε, στη δική μας νομοθεσία. Γι' αυτό ακριβώς θα εργαστούμε προκειμένου οι εργασίες εξέλιξης του ενεργειακού πακέτου και των κλιματικών αλλαγών να ε, είναι επιτυχής. Θα συνεχίσουμε επίσης να εργαζόμεθα για το νομοθετικό πλαίσιο σε θέματα αποτελεσματικότητας της ατμόσφαιρας και του ε, βιομηχανικού περιβάλλοντος, καθώς επίσης και τις διεθνείς συμβάσεις μίζουν τα θέματα αυτά. Θα θέλαμε να διατηρήσουμε τον ηγετικό ρόλο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μείωση και στην εξάλληψη των ε, ρηπογόνων εκπομπών, όπως επίσης και την βιώσιμη ανάπτυξη των ε, χημικών προϊόντων. Θέλουμε να έχουμε τις ελάχιστες δυνατές ε, επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και στην υγεία των πολιτών μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντική νομοθετική προσπάθεια σε θέματα χημικών ουσιών. Αναφέρομαι στον κανονισμό REACH ε, και ο οποίος αφορά όλες τις ε, χημικές ουσίες και όλους τους αντίστοιχους κανονισμούς που έχουμε για τις επικίνδυνες ουσίες η Ισπανία θα ήθελε να προχωρήσει την αναθεώρηση αρκετών ε, οδηγιών που σχετίζονται με τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κατάλοιπα για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο αποτελεσματική διαχείριση και να μειώσουμε τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον. Επιπλέον, θέλουμε να προωθήσουμε συγκεκριμένη νομοθεσία για την ανακύκλωση των βιοκαταλήπων. Το έδαφος είναι ιδιαίτερα ευάλωτο, πολύ σημαντικό για το περιβάλλον και τις ε, οικονομικές δραστηριότητες. Γι' αυτό ακριβώς το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να του δώσουμε την ίδια ευρωπαϊκή προσοχή που έχουμε δώσει στον, ε, στην ατμόσφαιρα, στον ατμοσφαιρικό αέρα και στο νερό. Ξέρουμε τι προσπάθειες έχουν κάνει κάποια κράτη-μέλη για να έχουμε μια κοινή απάντηση. Γνωρίζω ότι δεν θα είναι εύκολο, αλλά είμαι βέβαιη ότι θα μπορέσουμε από κοινού να καταλήξουμε σε συμφωνία για την ε, οδηγία για την προστασία του εδάφους. Όσον αφορά τώρα στην πρόταση κανονισμού για τις ε, μη εμπορικές ε, μετακινήσεις των οικώστων ζώων, των ζώων συντροφιά, πιστεύω ότι θα πλησιά, ε, πλησιάζουμε προς μια αίσια κατάληξη. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή ε, τον κανονισμό πριν από την 1η Ιουλίου, στην οποία 1η Ιουλίου λύγει και η μεταβατική περίοδος. Μια άλλη από τις πτυχές που θα θέλουμε να αφιερώσουμε το χρόνο μας είναι η απώλεια τη βιοπικιλότητας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θεωρούμε ότι αυτή είναι μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το 2010 είναι το Διεθνές Έτος Βιοπικιλότητας και γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε εις βάθος το θέμα αυτό αναλαμβάνοντας προκλήσεις και καθορίζοντας τους αντικειμενικούς μας στόχους για το 2010. Η Προεδρία μας επίσης είναι αρμόδια για την προετοιμασία της κοινοτικής συνεισφοράς στη διεθνή συζήτηση που θα γίνει στην Ιαπωνία στο δεύτερο εξάμεινο του 2010. Στην COP10 της ε, διάσκεψης της βιοπικιλότητας. Η ε, διάσκεψη για τη βιοπικιλότητα που θα γίνει στη Μαδρίτη, ένα φόρουμ συζήτησης ε, για την απώλεια βιοπικιλότητας, χρησιμοποιείται ως ε, ε, βάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προετοιμασία μας ε, για το συζήτηση που θα γίνει σε διεθνές επίπεδο. Ένα ακόμα από τα στοιχεία που θα θέλαμε να συζητήσουμε στη διάρκεια της Προεδρίας μας είναι η προστασία των δασών. Όπως ξέρετε η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγαλύτερη συχνότητα με φαινόμενα που πλήττουν τα δάση μας. Πυρκαγιές, πλημμύρες, όλα αυτά ευνοούνται από την αλλαγή του κλίματος. Τα φαινόμενα αυτά, τα οποία προκαλούν τεράστιες ζημίες ε, στην ε, δασική μας κληρονομιά και στη βιοπικιλότητα, δεν γνωρίζουν σύνορα. Η πράσινη βίβλος για την προστασία των δασών και των ε, συστημάτων δασικών πληροφοριών θα χρησιμοποιηθεί ως βάση από πλευράς κρατών μελών για την βιώσιμη προστασία των δασών. Επιπλέον, στη διάρκεια αυτού του εξαμήνου θα γίνει μια υπουργική διάσκεψη η οποία θα είναι αφορερωμένη στην προστασία των δασών και ε, για τα αποτελέσματα θα ε, τα παρουσιάσουμε για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος στις 21 21 Ιουνίου του 2010. Μία άλλη από τις προτεραιότητες που έχουμε σε θέματα περιβάλλοντος είναι η διαχείριση των υδάτων. Θεωρούμε ότι είναι ένα περιβαλλοντικό μεν στοιχείο, αλλά ταυτοχρόνως ένα οικονομικό και κοινωνικό στοιχείο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν απαντήσεις ε, στα ε, πολύ προβλέψιμα σενάρια που έχουμε για τις ε, τεράστιες πλημμύρες που θα προκύψουν από την αύξηση των θερμοκρασιών και τις πλημμύρες που θα προκύψουν και από τις κατακλυσμίες βροχοπτώσεις η Υπουργική Διάσκεψη για την ε, Μεσογειακή Στρατηγική Δάτων που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες της Μεσογείου θα είναι μια έξοχη δυνατότητα για να συζητήσουμε από κοινού ε, τα φαινόμενα αυτά και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, όπως επίσης και η Διεθνής Διάσκεψη για την ε, ξηρασία και την έλλειψη ύδατος που θα γίνει στις 28 και 29 Φεβρουαρίου. Προσπάθησα να σας δώσω συνοπτικά τους ε, στόχους που θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε στη διάρκεια της Προεδρίας μας. Όλοι αυτοί οι στόχοι είναι δυνατόν να υλοποιηθούν μόνο εάν η Προεδρία μας καταφέρει να ε, έχει και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάθε ενός από εσά εδώ στην Επιτροπή σας. Εγώ προσφέρω την ε, συνεργασία μου για να μπορέσουμε να πετύχουμε. Και εδώ ε, βρίσκομαι μεν σήμερα, αλλά θα είμαι διαθέσιμη όποτε με χρειαστείτε, προκειμένου να προσπαθήσουμε να συντονιστούμε, να ενώσουμε τις προσπάθειές μας και να καταφέρουμε να έχουμε μια Ευρώπη η οποία περιβαλλοντικά θα είναι πολύ πιο βιώσιμη, διότι δεν μπορούμε να αρνηθούμε κάτι τέτοιο στις μελλοντικέ γενοές Ευρω... ε... Ευρωπαίων ανδρών και γυναικών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Υπουργό κυρία Σπινόζα. Ε, πολύ αισιόδοξο πρόγραμμα. Σημείωσα 12 σημεία από αυτά τα οποία αναφέρατε. Μια ντουζίνα μέτρα λοιπόν τα οποία βρίσκονται στο πρόγραμμα της Ισπανικής Προεδρίας και θα απασχολήσουν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα συνεδριάζει και η Κορεπέρη, μόνιμη αντιπροσωπεία, για το θέμα του ε, τι θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως θέση της στα Ηνωμένα Έθνη για τις 31 Ιανουαρίου. Θα δούμε αν θα ισχύσει ε, το 2020 ή αν θα μπει κάπου και ο ρυθμός του 30. Ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να εκφράζεται με μία ενιαία φωνή για τα θέματα αυτά. Για το πρώτο θέμα που αναφέρεται, για την προστασία του κλίματος. Δίνω το λόγο στον Ρίχα Τζέμπερ καταρχήν. Και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι ομιλητέ. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο μου, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ και την Υπουργό. Ευχαριστούμε που ήρθατε και παρουσιάσατε το πρόγραμμα τη Ισπανική Προεδρία από αυτά τα οποία είπατε. Σημείωσα ότι είναι πολύ σημαντικά τα θέματα περιβάλλοντος και συνδέονται στενά με τα θέματα της οικονομίας. Και πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι είναι σημαντικό το θέμα της προστασία του κλίματος, αλλά γνωρίζετε κι εσείς ότι πολύ συχνά δεν ζητήθηκε η γνώμη μας και φάνηκε ότι δεν εκφράστηκε η Ευρώπη με μία φωνή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν τι σκοπεύετε να κάνετε ως Προεδρία, ούτως ώστε να εκφράζετε η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με σαφήνεια, με μία ενιαία θέση. Αυτή η έλλειψη ενότητας που υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών, πώς είναι δυνατόν να γεφυρωθεί αναφέρετε το θέμα της διαχείρισης των υδάτων και εσείς προέρχεστε από μια χώρα με πολύ ήλιο αλλά δυστυχώς με λίγους ε, υδατικούς πόρους και αναφέρατε ε, διάφορες διασκέψεις αλλά δεν είναι ε, ξεκάθαρο ποια είναι η θέση της Ισπανικής Προεδρίας πώς ε, ε, θα προωθήσετε την, ε, τις νομοθετικές διατάξεις για το νερό και την οδηγία για το νερό. τι γίνεται σε κάθε κράτο μέλο και στο δικό σα συγκεκριμένα κράτο μέλο. Γιατί ξέρουμε ότι η Ισπανία καταναλώνει σε μεγάλο βαθμό νερό για τη γεωργία. υπάρχει δυνατότητα χρήσης νέων τεχνικών από τους αγρότες, ώστε να μειώνεται η κατανάλωση ύδατος. Πώς θα αντιμετωπίσετε λοιπόν αυτό το βασικό ε, πρόβλημα και με ριζικό τρόπο. Επίσης, ε, τι πρωτοβουλίες μπορούν να δοθούν για την πρόθεση νέων τεχνολογιών, ε, για το σχεδιασμό προϊόντων, ούτως ώστε να αποφεύγεται η κατασπατάληση των υδατικών ε, πόρων και για να μπορέσουμε να έχουμε σωστή διαχείριση στο μέλλον. Ένα επόμενο σημείο όσον αφορά ε, την ε, οδηγία IPPC θέλουμε να έχουμε ε, ως το δυνατόν ενιαία πρότυπα στην Ευρώπη και ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη ε, ε, ανομοιογένεια των απόψεων στο Συμβούλιο Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και διαφορετικά μέτρα αντιμετώπισης. Ποιες είναι οι προθέσεις σας λοιπόν για αυτό το θέμα, ούτως ώστε να γεφυρώσετε τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν. Και όταν μιλάτε ε, για τα ε, ε, απόβλητα, ελπίζω ότι θα τηρήσετε αυτό το οποίο είπατε, ότι θα καταλήξετε σε κάποια σημαντική πρόταση για αυτό το τομέα. Ευχαριστούμε πολύ τον Ιχατζέμπερ. Έχω 20 αγορητές και κλείνω τώρα τον κατάλογο των αγορητών. Δεν το λόγο στη Λίντα. Καλό θα ήταν να είχαν οι συντονιστέ 2,5 λεπτά για να προλαβαίναμε καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη, λέει, κυρία Μακάβαν. Καλώ ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Τα είπαμε και στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα. Το θέμα στο οποίο θέλω να εστιάσω την προσοχή μα ε, είναι η Κοπεχάγη και το τι θα συμβεί μετά την Κοπεχάγη. Νομίζω ότι δεν είμαι η μόνη που έχει μπερδευτεί για το τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Την περασμένη εβδομάδα ο Ιβο Ντεμπόρ ανακοίνωσε, από ό,τι κατάλαβα εγώ, τις 31 Ιανουαρίου, τα διάφορα μέρη ε, που σημείωσαν τη συμφωνία της Κοπεχάγης ε, θα υποβάλουν τα σχέδια εκπομπών τους στα Ηνωμένα Έθνη. Την περασμένη εβδομάδα ακούσαμε ότι είναι κάπως ευέλικτη αυτή η ημερομηνία του τέλους Ιανουαρίου. Εσείς, Υπουργοί Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, πώς το βλέπετε, πώς θα παρουσιάσουμε εμείς τα δικά μας στοιχεία γιατί άκουσα επίση ότι η Γαλλία θα υποβάλει διαφορετικά στοιχεία σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα έχουμε λοιπόν ενιαία στοιχεία που θα δώσουμε στα Ηνωμένα Έθνη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Άνοιξη επικείται και αυτή η συνάντηση στη Βόνη. Πώ θα προετοιμαστείτε για τη Βόνη. Και ε, πώς θα ανακτήσουμε την όθηση και τον ενθουσιασμό που υπήρχε ε, με την προοπτική της συνάντησης στο Μεξικό και φαίνεται ότι ο Ομπάμα άλλαξε την προτεραιότητα, σαν να περνάει από την αλλαγή του κλίματος πάλι στα θέματα της οικονομίας. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτό το οποίο θέλουμε θα γίνει τελικά. Ευχαριστώ. Chris Davis. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, ε, έχουμε μια κρίσιμη συνάντηση της ε, Επιτροπή για το Κλίμα την επόμενη Τρίτη και θέλω να ακούσω τι κάνει η Προεδρία για να εξασφαλίσει τη θετική έκβαση της συνάντηση. Και θα ήθελα να πω προς του συναδέλφου ότι πριν από τρία χρόνια αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχουμε μέχρι το 2015 προγράμματα για την ε, δέσμευση και αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακος. Δεν έδωσε όμως τα κονδύλια που θα χρησιμεύαν για την τεχνολογία αυτή. Και ε, τώρα λέμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε κονδύλια από το ε, πρόγραμμα ανταλλαγή εκπομπών διευθύντου του άνθρακο, αλλά έχει περάσει πάνω από ένα χρόνο από τότε που αποφασίστηκε και δεν έχει γίνει τίποτα από αυτού. Έχουμε λοιπόν αφήσει ένα χρόνο να περάσει χωρί να κάνουμε τίποτα. Και η Επιτροπή ε, προετοιμάζει μια, έχει προετοιμάσει μια απόφαση που θα συζητηθεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντο την επόμενη ε, εβδομάδα σχετικά με τα διάφορα προγράμματα για ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια ή για το πρόγραμμα CCS και κάνει και μια κατανομή τη χρηματοδότηση. Έχει υποβληθεί και μια εναλλακτική πρόταση Τράπεζα από τη Γερμανία προσπαθεί να επανεθνικοποιήσει τη χρηματοδότηση. Λέει δηλαδή να η χρηματοδότηση α τη μοιράσουμε μεταξύ 27 κρατών μελών. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ποτέ δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Καλύτερα να αποσύρουμε ολόκληρο το πακέτο παρά να έχουμε ε, κάτι σε εθνικό επίπεδο για αυτά τα προγράμματα επίδειξη. Στην αρχή της εβδομάδας ε, φαίνονται, ε, τα σημεία, φαίνονται αμφίσιμα τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο Συμβούλιο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην ψηφοφορία. Συνεχίζουμε να ζητάμε ε, ένα μέλλον ε, με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρωπος. Επομένως, τι κάνει το Συμβούλιο για να έχει θετική έκβαση στη ψηφοφορία αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Σαμχήν Μπελιέ. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας. Η Ισπανική Προεδρία έχει βάλει στο πρόγραμμά της ε, την νομοθεσία για την προστασία του εδάφους πολύ καλό αυτό το σημείο. Άλλο ένα θετικό σημείο είναι ότι αποφασίσατε από ό,τι φαίνεται να ξαναρχίσουν οι εργασίες στο Συμβούλιο με βάση το κείμενο που απολύθηκε επί Πορτογαλικής Προεδρίας το 2007, ένα κείμενο το οποίο κατά τη γνώμη μας ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσει, αλλά χώρε μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο διαφωνούν με το πρόγραμμα, με το σχέδιο οδηγίας, διότι το θεωρούν πολύ δεσμευτικό και πολύ απαιτητικό. Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι συμφωνούμε ότι είναι απαραίτητο να έχουμε κοινού κανόνε για το έδαφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά ε, τη ρήπανση του εδάφου για την διατήρηση του πλούτου ε, των εδαφών μας και για να εγγυηθούμε την ποιότητα των υδάτων, την ποιότητα της γεωργικής παραγωγής, τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς καθώς και της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών. Κύριε Υπουργέ, έναντι της ε, ε, μειοψηφία, της ανασταλτικής μειοψηφίας στο Συμβούλιο. Νομίζω ότι θα υπάρχει κάποια συμφωνία μέχρι τις 15 Μαρτίου το αργότερο και επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο είναι έτοιμη η Ισπανική Προεδρία να κάνει συμβιβασμού και ποια είναι τα όρια, πού βάζετε την κόκκινη γραμμή πέρα από την οποία δεν θέλετε να φτάσετε στην αναζήτηση συμβιβαστικών λύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Εγώ εκπλήσωμαι που το πρόγραμμά σας εστιάζει απλώς και μόνο σε περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία σχετίζονται είτε με την αποτυχία του COP15 είτε με την προετοιμασία του COP16. Όταν συζητήθηκε το θέμα της μεγάλης ρήπανσης, ποια ήταν οι βιομηχανίες που ε, μόλυναν, που ρήπαιναν το περιβάλλον. Όταν ε, μιλούσαμε για πράσινη γη, ήταν πράσινη γη. Τότε ποιος ήταν αυτός ο οποίος ε, ρήπαινε το περιβάλλον. Ως υπουργό Περιβάλλοντος θα πρέπει να ασχολείστε με τα πάντα και με το COP16, αλλά θα ήθελα να ξέρω και τι γίνεται η θέση σας ε, για τις μεγάλες ε, περιβαλλοντικές προκλήσεις οι οποίες δεν τηρούνται. τα απορρίμματα στη θάλασσα. Ξέρουμε ότι η θάλασσα θάλασσές μας είναι γεμάτες από απόβλητα. Τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό. Και τι θα γίνει και με προϊόντα τα οποία εισάγονται όλο ένα και περισσότερα από τρίτες χώρες οι οποίες ε, ρηπαίνουν. Ε, ή τι γίνεται με τα φυτοϊγειονομικά προϊόντα, τα διάφορα φυτοφάρμακα και παρασιτοκτόνα που απαγορεύονται αλλά κυκλοφορούν ελεύθερα στα τραπέζια μας, ναι. πάνε στα παιχνίδια των παιδιών μας και πολύ τακτικά βρίσκονται και σε προϊόντα τα οποία υπόκεινται πέραν επεξεργασία. Τι άποψη έχετε για τα πυρηνικά, για την διαχείριση των ε, πυρηνικών αποβλήτων. Ε, τι γίνεται με την ε, οδικέ, οδικές μεταφορές, τις σιδηροδρομικές μεταφορές οι οποίες ρηπαίνουν και σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. τι σκοπεύετε να κάνετε για να δώσετε κινήτρα σε χώρες οι οποίες παράγουν ενέργεια και δεν ε, κοιτούν ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκή, ε, ηλιακή ενέργεια. Εγώ θα ήθελα να κατανοήσω όλα αυτά τα πράγματα από το πρόγραμμά σας. Δεν υπάρχουν μόνο τα θέματα που σχετίζονται με την αλλαγή του πλα, κλίματος. Έχουμε και όλα τα υπόλοιπα. Το περιβάλλον είναι ένα αμάλγαμα πραγμάτων. Πέστε μας κάτι. Ευχαριστούμε. Η Κρίστα Κλάς παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρεύουσα του Συμβουλίου θα μπορούσα άμεσα να συνεχίσω αυτά που είπε ο συνάδελφο Ρώση. Και εγώ βλέπω να λείπουν τα πρακτικά χειροπιαστά πράγματα που το επόμενο εξάμεινο η Ισπανική Προεδρία θέλει να αναλάβει και όπου βρισκόμαστε μπροστά σε νέε αποφάσεις. Και τώρα σε σχέση με αυτό το οποίο είπατε και για το έδαφος. Στην ίδια γραμμή τοποθετηθήκατε όπως για τον ατμοσφαιρικό αέρα και το νερό. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Είναι διασυνοριακά ε, στοιχεία ο αέρας, ο ατμοσφαιρικός ε, και το νερό. Όμως ε, το έδαφος έχει όρια. Πρέπει να δεχθούμε ότι εδώ έχουν ειδικέ υποχρεώσεις τα κράτη-μέλη για τη διαφύλαξη των εδαφών, της γης, του εδάφους και όταν έχουμε και την προστασία του εδάφους σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει πρέπει να δούμε ξεχωριστά αυτό το θέμα. Επίσης το θέμα για τα βιοκτώνα και τον κανονισμό. Είπατε τα οικοσυστήματα και η υγεία των πολιτών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να προστατεύονται. Τι θα κάνει λοιπόν η Ισπανική Προεδρία όσον αφορά τον κανονισμό για τα βιοκτώνα που έχουμε μπροστά μας. Θα ασκήσετε πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρχει μια μελέτη επιπτώσεων, impact assessment, γιατί πρέπει να αποτιμήσουμε, να αξιολογήσουμε ποια ε, στοιχεία είναι εκείνα τα οποία ε, είναι ιδιαίτερα ε, σημαντικά, επιβαρυντικά για την υγεία. Έχουμε και το καθήκον προστασίας της υγείας ε, και των υγειονομικών διατάξεων. Τι πρέπει να γίνει. Και εδώ το στενότερο πλαίσιο το, στο οποίο έχουν διατυπωθεί θα θέλαμε να εξεταστεί από την Ισπανική Προεδρία, να υπάρξει μια τοποθέτηση. Πώς αντιμετωπίζει η Ισπανία το θέμα, το ότι περισσότερα θα θέλαμε να μεταφερθούν στο ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την αδειοδότηση, όσον αφορά αυτά τα, αυτές τις ουσίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κλάση είναι η συγγήτρια για τα βιοκτώνα. Ο Κρήτον Αρσένης παρακαλώ έχει τον λόγο. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, Υπουργέ. Σας ε, ε, καλωσορίζουμε και το θέμα της βιοπικιλότητας, ε, διότι η προστασία της βιοπικιλότητας πρέπει να δούμε πώς θα συνδέεται με την προστασία των οικοσυστημάτων και που τώρα βλέπουμε ότι 50% σε σχέση με τις εκπομπές ρήπων αυτές αφομοιώνονται από πλευρά των ε, δασών και των οικοσυστήματων. Υπήρχε η πρόταση καθορισμού των ε, ε, όσων γίνονται από εκείνου που αποψηλώνουν τα δάση και διαθέτουν την ξυλία στις ευρωπαϊκές αγορές. Θα πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα ξεχωριστά. Υπάρχει και απογοήτευση από πολλούς σε σχέση με αυτό. Από ό,τι φαίνεται δεν απαγορεύεται η παράνομη διάθεση, η διάθεση παράνομης ξυλίας στις ευρωπαϊκές αγορές. Τι θα γίνει σε σχέση με την εποπτεία. Θα παραμείνουν τα θέματα αυτά στους ίδιους, ε, στις ίδιες επιχειρήσεις που αποψηλώνουν τα δάση. Και όσον αφορά και το ποσοστό των ε, ε, εκπομπών ρήπων, κάποιοι λένε ότι αν απαγορευόταν η παράνομη ξυλία στην ευρωπαϊκή αγορά, θα είχαμε μια σαφή υποχρέωση επιπλέον για το στόχο, επί, του στόχου ε, του 2020 σε στόχους. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Ισπανικής Προεδρίας. Ποια συνέχεια θα δοθεί σε σχέση με τα θέματα αυτού του κανονισμού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. <coughs> Κέβιν Άντι παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι ευχαριστώ την Ισπανίδα Υπουργό για το ότι ήρθε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Είναι δύσκολη η χρονική στιγμή κατά την οποία αναλαμβάνει την πρωτοκαθεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω όσον αφορά την βιοπικιλότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Έχετε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ως Ισπανική Προεδρία και θέλω να σας συγχαρώ γι' αυτό. Θέλω να επικεντρωθώ στην βιοπικιλότητα. Αναφερθήκατε σαν μία από τι μεγαλύτερες προτεραιότητες σε σχέση με την προστασία της βιοπικιλότητας. Επίσης αναφέρατε τα θέματα της προστασίας των δασών και της βιοπικιλότητας ε, στους ωκεανούς, ε, στη θάλασσα. Θέλω να σας πω ότι σήμερα ψηφίσαμε θέματα site στην Επιτροπή μας, προστασίας ειδών υπό εξάλληψη, που απειλούνται με εξάλληψη και είμαστε υπέρ της ε, απαγόρευσης της απεριόριστης αλληλείας του τόνου. Τι κάνετε σχετικά, μια και είναι γνωστό ότι υπάρχει προσπάθεια να απαγορευτεί αυτή η αλληλεία Ιταλία και από τους Ιταλούς και στη Γαλλία επίσης υπάρχει ένα μέτωπο μεσογειακών χωρών όσον αφορά την απαγόρευση αλίας και εδώ θα έπρεπε να το δούμε αυτό το θέμα και να δούμε ποιο ρόλο θα διαδραματίσετε εσείς επίσης για την απαγόρευση της ε, εμπορίας ελεφαντοστού μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την Υπουργό που ήρθε σήμερα. Σας ευχαριστώ γιατί μας παρουσιάσατε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα. Κάποιοι συνάδελφοι ήδη μίλησαν για το θέμα του μετά την Κοπεχάγη. Εγώ θα άρχισα να το αποκαλώ πριν από το Μεξικό, γιατί μας ενδιαφέρει το πώς θα έχουμε καλύτερη εμφάνιση στο Μεξικό ως Ευρώπη. Και εδώ θα ήθελα να είναι πιο κριτικές οι παρατηρήσεις μου. Μέχρι τώρα μιλάμε για τη βελτίωση του ρόλου της Ευρώπης, αλλά αυτό το οποίο δεν βλέπω να υπάρχει είναι ότι δεν φαίνεται να τονίζουμε τον επίγοντα χαρακτήρα. Ήδη πρέπει να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα. Και δεν ακούω και πολύ συγκεκριμένα προγράμματα από την Ισπανική Προεδρία για το πώ θα βελτιώσει το ρόλο τη Ευρώπη. Και αν δείτε τη συζήτηση που γίνεται για το 20%-30%, φαίνεται ότι ε, στο παράδειγμα φαίνεται ότι η Ευρώπη δεν έχει διδαχθεί από τα λάθη τη. Την ίδια συζήτηση ξανακάνουμε. Πολύ συγκεκριμένα λοιπόν αυτά τα ερωτήματα που έχω για την Ισπανική Προεδρία. Πρώτον, συμφωνούμε όλοι ότι η Ευρώπη θα πρέπει να εκφράζεται με ενιαία φωνή και αυτό να γίνει και στο Μεξικό, αλλά ποιο θα μιλήσει με την ενιαία αυτή φωνή και η Ισπανική Προεδρία ποιο πιστεύει ότι θα πρέπει να μιλήσει με αυτήν μια ευρωπαϊκή φωνή. Και δεύτερον, την περασμένη εβδομάδα οι βασικές χώρες είπαν ότι θέλουν να γίνει ήδη το Μάρτιο κάποια συνάντηση στα Ηνωμένα Έθνη. Καλή ιδέα είναι αυτό, αλλά ε, πήγε η Ευρώπη και είπε σε αυτές τις χώρες ε, συμφωνούμε μαζί σας και θέλουμε να συνεργαστούμε και να είμαστε μαζί σας σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Έχει πάρει πρωτοβουλίες ε, η Ισπανική Προεδρία ώστε να μπει η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτές τις βασικές χώρες το Μάρτιο στη συνάντηση. Ευχαριστώ. Νίκ Γκρίφιν. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Υπουργέ, χτε τρει Γερμανοί ε, επιστήμονε για το κλίμα έγραψαν στο Σπίγκελ ένα άρθρο ιδιαίτερα ε, επικριτικό όσον αφορά την αλλαγή του κλίματο, όχι μόνο για τους πάγου στα Ιμαλάια, αλλά και για άλλες εκθέσεις που βασίζονται σε άρθρα που δεν, είναι, δεν έχουν αξιολογηθεί από ομοτήμους. Το ένα αφορά αυτό που είπατε και εσείς στην αρχική σας ε, ομιλία σχετικά με τη σύνδεση των ε, πυρκαγιών στα δάση με την αλλαγή του κλίματος. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, με επιστημονικά δεδομένα. Θα αναλάβει ε, η Ισπανική Προεδρία κάποια επανεξέταση των εσφαλμένων επιστημονικών στοιχείων. Πόσα στοιχεία θέλετε για να πιστείτε να το κάνετε. Δεύτερον, έχω λάβει επιστολές από Βρετανούς που ζουν ζουν στην Ισπανία και μερικέ φορέ και συγκλονιστικά γράμματα. Ένα, σπίτι, ε, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ε, που καταστράφηκε το σπίτι του σύμφωνα λόγω τη νομοθεσία του 88 και σύμφωνα με την έκθεση ΟΚΕΝ θα έπρεπε η Ισπανία να σταματήσει να εφαρμόζει αυτό το νόμο. Δεν τηρούνται όμω αυτέ ε, οι διατάξει. και νομίζω ότι είναι παράδοξο το ότι αγνοείται η θέση του Κοινοβουλίου από την Ισπανική κυβέρνηση με τα μέτρα τα οποία ακολουθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε ήδη τις πρώτες δέκα ερωτήσεις μπορεί να απαντήσει η κυρία Υπουργό για το ΣΑΙΤΕΣ, για την αλλαγή του κλίματος, για τη βιοπικιλότητα, για το έδαφος. Αν θέλετε να λάβετε το λόγο για να απαντήσετε στις πρώτες, στο πρώτο γύρο ερωτήσεων, κύριε Υπουργέ. Eh, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε θα απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις επιχειρώντας ταυτόχρονα να δώσω και περισσότερες πληροφορίες από αυτές που σας έδωσα στην πρώτη παρέμβαση μου. Ο κύριος Σέμπερ μας έθεσε το θέμα της Κοπενχάγης. Αναγνωρίζω ότι ήμουν λίγο λακωνική στην πρώτη μου παρέμβαση, αλλά σας είχα πει ότι Ήμουν στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα, γι' αυτό προσπάθησα να διαφοροποιήσω λίγο την παρέμβασή μου. Τι πρέπει να κάνουμε μετά από την Κοπενχάγη, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε ε, ως Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Προεδρία. Από πλευράς Προεδρίας δεν μπορούμε να πέσουμε σε μελαγχολία. Δεν μπορούμε να βλέπουμε στην Κοπεχάγη όλα όσα δεν έγιναν και θα μπορούσαν να είχαν συμβεί. Θα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, όπως έλεγε και ο κύριος Έικχουτ, και να κοιτάμε ήδη μπροστά στο Μεξικό. Το να κοιτάμε λοιπόν προς το Μεξικό σημαίνει ότι θα πρέπει να εργαστούμε σε δύο τομείς. Σε διεθνές πλαίσιο προκειμένου η Ευρώπη να συνεχίσει να έχει τον ηγετικό της ρόλο και για να μπορέσουμε να επιτύχουμε όταν θα φτάσουμε στο Μεξικό στα τέλη αυτού του εξαμήνου να είναι πολύ πιο πάγια η θέση μας διεθνώς και να μην υπάρχουν οι αποκλήσεις που είχαμε μέχρι τούδε. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει μια τεράστια προσπάθεια και η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει από την Ευρώπη όπως γινόταν και στο παρελθόν διότι η Ευρώπη πάντα ήταν ηγέτης. Χάρη στην Ευρώπη καταφέραμε να καταλήξουμε σε όλα όσα ε, καταλήξαμε στην Κοπεχάγη και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Εάν δεν ήταν ο κοινό μας ρόλος η Κοπεχάγη σίγουρα θα ήταν μια τεράστια αποτυχία. Ε, ενώ μιλούσαμε υπήρχε μια συνεδρίαση στην Κορεπέρ μόλις μου έδωσαν και το σημείωμα ε, ζητώ συγγνώμη επειδή μόλις μου το δώσανε θα σας το διαβάσω αυτό Η Κορεπέρ μόλις κατέληξε σε συμφωνία πριν από λίγα λεπτά ε, στην αποστολή επιστολής από πλευράς Προεδρίας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να επιβεβαιώσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται με τη Συμφωνία της Κοπενχάγης και για να επιβεβαιώσει και τις δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ανεξάρτητος στόχος της τάξης του 20% και ε, δεσμευμένος στόχος του 30%. Αυτό είναι λοιπόν η συμφωνία που μόλις υιοθετήθηκε ομόφωνα και αυτό επιβεβαιώνει ότι θα μιλάμε και πάλι με μία φωνή. σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να επικεντρωθούμε όχι μόνο στις Ηνωμένε Πολιτείε, όπως ε, θεωρούν κάποιοι, ε, ξέρω ότι δεν το πιστεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά όπως πιστεύουν κάποιοι, θα πρέπει όμως να κάνουμε και μια μεγάλη προσπάθεια με αναδυόμενες χώρες και με χώρες ε, υποανάπτυξη. Μπορούμε να το κάνουμε και εγώ θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να καθυστερήσουμε ούτε ένα λεπτό ε, παραπάνω ε, γιατί στο Μεξικό, στο Μεξικό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε τη συμφωνία που θέλουμε όλοι. Μία συμφωνία που θα είναι δεσμευτική και που θα μας οδηγήσει σε μείωση εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο γιατί το να συζητούμε την αλλαγή του κλίματος ε, το ξέρετε καλύτερα από μένα δεν είναι μόνο η Ευρώπη, δεν είναι μόνο ε, κάθε ένα από τα 27 κράτη-μέλη αλλά είναι μία παγκόσμια πολιτική και μια πολιτική για την οποία θα πρέπει να δεσμευτούμε όλοι, πολίτες, θεσμικά όργανα και κυβερνήσεις, προκειμένου να επιτύχουμε το στόχο που επιθυμούμε όλοι. Ο πλανήτης μας να χρησιμοποιεί λιγότερο άνθρακα και κατά συνέπεια να έχει λιγότερες εκπομπές. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον πλανήτη μας για το μέλλον. Ένα Άλλο θέμα το οποίο έθεσε ο κύριος Σέιμπερ ήταν ε, οι στόχοι για το νερό. Το να μιλάμε για το είδωρ είναι ε, μια συζήτηση που ε, αφορά ένα αγαθό το οποίο είναι όλο και σπανιότερο ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία διαμένουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι υπάρχουν χώρες που πλήττονται περισσότερο από την έλλειψη ύδατος και κάποιες άλλες έχουν ήδη πληχτεί ή θα μπορούσαν να πληγούν στο μέλλον όχι όμως μόνο από την έλλειψη νερού ως αγαθό, αλλά και από τα ακραία φαινόμενα που εκδηλώνονται ε, όλο και περισσότερο συχνά. Μπορεί να υπάρξει μια εβδομάδα εξαιρετικής ξηρασίας και την επόμενη εβδομάδα στην ίδια περιοχή της Ευρώπης η ίδια περιοχή να ε, πλημμυρίσει. Προσπαθούμε λοιπόν να μην ε, εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα και αν εμφανίζονται να προκαλούν όσο το δυνατόν λιγότερες ζημίες. Πώς μπορούμε να μειώσουμε την έλλειψη νερού. Νομίζω ότι από πλευράς Προεδρίας υπάρχουν δύο θέματα τα οποία θα πρέπει να προωθήσουμε. Αφενός ε, να επιτύχουμε μείωση από όλε τις ε, πλευρές, από την καθημερινή χρήση των πολιτών, το πώ χρησιμοποιούμε νερό όλοι μας, όπως και όλες τις οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες γίνονται σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αλλά ταυτόχρονα εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες. Νέες τεχνολογίες οι οποίες μας επιτρέπουν να ανακυκλώνουμε νερό, αφού έχει ε, περάσει υποστή κατάλληλο καθαρισμό, βιολογικό καθαρισμό να ε, επαναχρησιμοποιείται, όπως επίσης αφαλατωμένο νερό, διότι μιλάμε για πόρους οι οποίοι δεν ε, ε, είναι σε έλλειψη. Επίσης, χρήση νέας ε, τεχνολογίας για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, βιομηχανικές περιπτώσεις και όλα αυτά θα πρέπει να αποτελούν ένα τέλειο κύκλο για να έχουμε ποιότητα στο νερό μας. Παραδείγματο χάρη, ε, ας πάρουμε μία πόλη, δεν μας ενδιαφέρει σε ποια χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, μία πόλη ε, που έχει τουριστική κίνηση και συνήθως αυτή η τουριστική κίνηση εμφανίζεται σε καλοκαιρινές περιόδους, σε περιόδους διακοπών. Εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση σε νερό από ό,τι θα μπορούσε να υπάρχει σε κάποια άλλη εποχή του χρόνου. Εάν το νερό που χρησιμοποιείτε υπόκειται καθαρισμό και από εκεί και πέρα ανακυκλώνεται, θα μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε για να διατηρηθεί ίσως μια ισορροπία στην ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται και που ε, ε, πλέον σήμερα ευτυχώς μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό λοιπόν είναι το σκεπτικό μας σε θέματα υδάτων. Και εδώ δεν θα πρέπει να λησμονούμε και μία σειρά από παράγοντες που μπορεί να ε, φαίνονται πολύ πιο συγκεκριμένοι, αλλά έχουν πολύ σημαντική επιρροή όπως είναι για παράδειγμα όλα τα θέματα της ε, αναδάσωσης των ε, ε, ορεινών μας εκτάσεων ή ότι ότι μπορούμε να κάνουμε με τις όχθες όλων των ευρωπαϊκών ποταμών. Υπάρχουν ακραία φαινόμενα. Τα ακραία αυτά φαινόμενα και το ανέφερα στην παρέμβασή μου. Θέλουμε να εργαστούμε με τέτοιο τρόπο αφενός ώστε να αποφύγουμε τις επιπτώσεις αν υπάρχουν τέτοιες ε, λειψιδρίες ε, ή αν έχουμε προβλήματα πλημμυρών. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό με προγράμματα για την αντιμετώπιση λειψιδρίας και ξηρασίας που έχουν κάποια ευρωπαϊκά κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη σήμερα. Αλλά πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να επεξεργαστούμε τέτοια σχέδια. Καθώς επίσης και την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρών στις ε, περιοχές που αντιμετωπίζουν τέτοιους κινδύνους και αυτό μέσα στο πλαίσιο των υδάτινων πόρων πρέπει να γίνει. κάποιες χώρες έχουν κάνει ήδη κάποια πράγματα, μπορούμε να κάνουμε μια πρόσθετη προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να βελτιώσουμε και να προετοιμαστούμε και μέσα στην οδηγία για το νερό, για τους υδάτινους πόρους να το κάνουμε. Αυτά πρέπει να γίνουν. Είναι θέματα που η ανάπτυξή τους είναι περίπλοκη και σύνθετη και όλα όσα θα μπορέσουμε να κερδίσουμε από αυτά είναι θέματα που θα πρέπει συνενετικά να προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε ώστε να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε, βελτιώσουμε ή προσαρμόσουμε ανάλογα με το πώς επιθυμείτε να το δείτε αυτό το θέμα, τα θέματα της οδηγίας πλαισίου από πλευράς Μακάβαν αναφέρθηκε, ρωτήθηκε τι αποφασίστηκε από πλευράς του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν η Γαλλία είχε υποβάλει κάποια διαφορετικά στοιχεία. Επαναλαμβάνω εγώ αυτό το οποίο μόλις σας διάβασα, αυτό λεξί, σε σχέση με τη συμφωνία της Κορεπέρ διότι αυτή η συνεδρίαση γινόταν ενώ ε, βρισκόμαστε εμείς σε αυτή την αίθουσα. Νομίζω σε σχέση με την ανησυχία σας στην οποία συμμεριζόμαστε μπορούμε να πούμε ότι ανήκει στο παρελθόν πια ανήκει στην ιστορία. Ξεπεράσαμε αυτό το πρόβλημα, περνάμε σε μια νέα φάση και ελπίζω ότι θα συμμεριστείτε μαζί μου το ότι είμαστε ενωμένοι και ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι στην πορεία όσον αφορά το μέλλον. Ο κύριος Ντέιβις επίσης σχολίασε σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές τα προγράμματα σύλληψης ε, ε, του άνθρακα και αποθήκευσης του άνθρακα εδώ κάνουμε λόγο για μια μελλοντική δυνατότητα ως προοπτική υπό το πρίσμα φυσικά της Ισπανικής Προεδρίας με μεγάλο μέλλον. Ένα μεγάλο στίχημα ευρωπαϊκό για την τεχνολογία, για την αποθήκευση και σύλληψη του άνθρακα. Και είναι αυτονόητο ότι όλοι μας θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ευδοκιμήσει, να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Έχουν κάποιες χώρες αποφασίσει ήδη την τοποθέτηση αυτών των αποθηκών και των στοιχείων και συγκεκριμένα προγράμματα τα πιλωτικά έχουν ξεκινήσει να σχεδιάζονται. Σίγουρα αληθεύει σήμερα ότι κανένας από εμά που βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα δεν θα μπορούσε κατά 100% να επικυρώσει απόλυτα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να επιτύχουν ή να προβλέψει τι θα μπορούσαν να πετύχουν αυτά τα σχέδια. Είναι όμως ένα μεγάλο ευρωπαϊκό στίχημα. Ένα μεγάλο ευρωπαϊκό στίχημα που μπορούμε να συμμεριστούμε και με άλλες χώρες. Και είναι φυσικό και αυτονόητο ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την πορεία προς αυτή την κατεύθυνση. Χωρίς να ξεχνάμε βέβαια αυτά τα οποία συνεπάγεται η επένδυση στην ανάπτυξη και στην καινοτομία. Διότι όλοι μας εδώ, αν μπορούμε πραγματικά να αν σκεφτόμαστε πριν από 20 χρόνια αυτά τα πράγματα δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε επικοινωνία με ηλεκτρονικά μηνύματα, με emails. Πριν από 20 χρόνια είχαμε fax τα οποία στέλναμε ο ένας τον άλλον και το θεωρούσαμε και προηγμένο αυτό. Το ίδιο πρέπει να θεωρούμε και για προγράμματα ανώτατης χρήσης τεχνολογίας, τεχνολογικά, όπως την σύλληψη και αποθήκευση άνθρακα. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε λοιπόν αυτή την πτυχή, ότι κάθε μέρα θα πρέπει να βελτιωθούν, να βελτιώνονται αυτές οι πτυχές, ώστε στο ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα όσο περνάει από το χέρι μας. Άλλος ε, ευρωβουλευτής έκανε λόγο για τα μολυσμένα εδάφη. Εγώ στη δική μου παρέμβαση προσπαθούσα να σας ε, διαβιβάσω το μήνυμα ότι είχαμε και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν δυσκολίες που αντιμετωπίζονται από πλευράς κάποιων κρατών μελών. Όμως αυτό δεν σημαίνει και δεν συνεπάγεται ότι καταβάλαμε την τελευταία ίστατη προσπάθεια. Η κοινοτική πολιτική για την προστασία των δαφών αποτέλεσε αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν ξεκίνησε η πρώτη προετοιμασία εγγράφων εργασίας. Η Ισπανία όταν δεν είμαστε ακόμα προεδρία και όταν δεν είμαστε μέλος ακόμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ε, δώσαμε όταν γίναμε μέλος ιδιαίτερη προσοχή και σε αυτό το πακέτο μέτρων, ρυθμιστικών μέτρων και προσπαθήσαμε να αποτροχοπεδηθεί, να προχωρήσει. Η προσπάθειά μας σήμερα που είμαστε Προεδρία πρέπει να είναι ακόμα μεγαλύτερη ακόμα. Και πράγματι απόψε θα διαξαχθεί μια συνάντηση ε, εργασίας τεχνικού χαρακτήρα με κάποια από τα κράτη-μέλη που έχουν συγκεκριμένες δυσκολίες για την προστασία των εδαφών. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να εξετάζουμε κάθε μία και όλες τις δυσκολίες που έχουν τα κράτη αυτά για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους. Το κάναμε με τον ατμοσφαιρικό αέρα, το κάναμε με ε, την ηχητική όχληση. Γιατί να μην μπορέσουμε να το κάνουμε και με τα εδάφη, την προστασία των εδαφών. Είναι στο χέρι μας μια μεγαλύτερη προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί και με τη μεγαλύτερη προσπάθεια, μεγαλύτερη προσπάθεια για διάλογο και συνένεση και έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε καλύτερα. Ο κύριος Ρώση επίσης έκανε μια αναφορά στις βιομηχανίες που μολύνουν, που ρηπαίνουν όσον αφορά επίσης και με τις μεταφορές, οδικές μεταφορές ε, και τι μπορεί να γίνει σε σχέση με φωτοβολταϊκές ε, παραγωγές. Ε, αν μπορούσαμε να αναφέρουμε όλα τα inputs για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε περιβαλλοντικά την Ευρώπη ή τι μπορεί να γίνει ώστε να βελτιωθεί η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, θα βλέπαμε ότι είναι απειράριθμες αυτές οι δυνατότητες και εναλλακτικέ δυνατότητες που έχουμε. Και θα ήταν ατέλειωτος ο χρόνος που θα χρειαζόταν για να συζητήσουμε λεπτομέρειες. Και εδώ και στην Ευρωβουλή έγινε λόγος και για τις ναυτιλιακές μεταφορές και για τις εναέριες μεταφορές και τις εκπομπές ρήπων που θα έπρεπε να ενταχθούν στους υπολογισμούς. Είναι μικρά βήματα που πρέπει να γίνουν και να συνεχιστούν. Για τις φωτοβολταϊκές ε, ε, δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Συμφωνώ μαζί σας. Μπορούμε να κάνουμε λόγο για ανανεώσιμες πηγές ενέργεια όπου ήδη στην Ευρώπη είμαστε πρωτοπόροι, προπομπή σε πολλές πτυχές από την παραγωγή ε, ανανεώσιμων ε, ε, πηγών ενέργειας. Και όχι μόνο μπορούμε να συνεισφέρουμε στην επίτευξη του 20% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μέλλον, αλλά αν συνεχίσουμε με το ρυθμό που έχουμε σήμερα, μπορούμε ακόμα παραπάνω να αυξήσουμε έτσι περαιτέρω αυτή τη συμμετοχή του 20% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Νομίζω με αυτόν τον τρόπο απαντώ, ανταποκρίνομαι κατά κάποιο τρόπο στην παρέμβαση της κυρίας Κλάς που έκανε λόγο για τον ατμοσφαιρικό αέρα, για το νερό και για την μεγάλη ευθύνη που έχουμε όλοι μας. Εμείς στην Ευρώπη, η Ευρώπη και κάθε ένα από τα κράτη-μέλη ξεχωριστά επίσης. Ο κύριος Αρσένης μας έκανε λόγο για την βιοπικιλότητα και την προστασία της. Εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα, θα επανέλθω και θα το σχολιάσω αμέσως στη συνέχεια. Έκανε λόγο λοιπόν για την βιοπικιλότητα. Και εγώ εδώ που και εγώ ε, με ταχύτητα γοργά είδα και παρουσίασα τα θέματα αυτά της Ισπανικής Προεδρίας εγώ θέλω να πω και να σας διαβιβάσω το μήνυμα για κάποιους από τους στόχους που έχουμε υπόψη να πετύχουμε στη δική μας Προεδρία, στη διάρκεια της. Πρώτον, ο θεσπισμός ενός συνολικού στόχου για την βιοπικιλότητα για την περίοδο μετά το 2010. Άλλος από τους στόχους μας είναι η αναθεώρηση του στρατηγικού προγράμματος ε, της ε, Συμφωνίας της Σύμβασης για την Προστασία της Βιοπικιλότητας. Ένας τρίτος άξονας η ολοκλήρωση των διεθνών διαπραγματεύσεων για την πρόσβαση στους ε, ε, πόρους αυτούς και την κατανομή ε, του ωφέλους όσον αφορά τις προσπάθειες. Και τέταρτον, τη θέσπιση μιας διεθνούς πλατφόρμας ώστε να μπορέσει να ενδυναμωθεί η αμφίδρομη δράση μεταξύ επιστήμης και πολιτικής όσον αφορά τα θέματα βιοπικιλότητας. Είναι ίσως ένα από τα θέματα τα οποία είναι πιο καινοτόμα που μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτά με αυτόν τον τρόπο. Και ένα πέμπτο θέμα, ίσως ο μεγάλος ξεχασμένος. Αλλά παρόλα αυτά γι' αυτό δεν είναι λιγότερο σημαντικό. Η βελτίωση της γνώσης για τις οικονομικές επιπτώσεις που υπάρχουν και που προκαλούνται από την απώλεια, καθημερινή απώλεια της βιοπικιλότητας. Ένα άλλο θέμα από τα όσα τέθηκαν σε σχέση με την βιοπικιλότητα και που πραγματικά έχω συνειδητοποιήσει για το ότι συζητήθηκε, για το ότι καλύφθηκε σήμερα από αυτή την ίδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή είναι η θέση σε σχέση με τον ερυθρόπτερο τόνο και θα ήθελα εδώ και το σάιτες να πω με κάθε σεβασμό για το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει επίσης ε, να συμβαίνει το ίδιο και έναντι του Συμβουλίου και έναντι και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να αναμείνουμε μέχρι ότου συντάξει και υποβάλει την αντίστοιχη πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δοθεί συνέχεια Νομίζω την πρόταση θα την έχουμε σε μια προθεσμία σχετικά ε, σύντομη και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες και τις προσπάθειες με τεκμήρια και ε, ε, προτάσεις που θα μας υποβληθούν για τη λήψη απόφασης πάντα με την αρχή της ομοφωνίας βέβαια, ομόφωνα. Ο κύριος Γκράφ μου είπε, έθεσε μια, έκανε μια παρέμβαση και για θέματα βιοπικιλότητας, περισσότερο συνδεδεμένα βέβαια με δασοπυρκαγιέ. Ίσως όμως εδώ μπορεί να μην εκφράστηκα πολύ σωστά. Δεν ήθελα να πω στην παρέμβασή μου ότι οι κλιματικές αλλαγές είναι εκείνες που προκαλούν περισσότερες δασοπυρκαγιές. Όχι. Εκείνο που ήθελα να σας διαβιβάσω ως μήνυμα είναι ότι σε ένα σημαντικό τμήμα της Ευρώπης πληττόμεθα από δασοπυρκαγιές ως μάστιγα. Αυτές οι δασοπυρκαγιές ε, μας οδηγούν σε μια απώλεια βιοπικιλότητας ε, σε πολύ σημαντικό βαθμό. Τα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν και αποδεικνύουν ότι πολλές από αυτές τις δασοπυρκαγιές συμβαίνουν στα ίδια τα δίκτυα Natura 2000, προστατευόμενες δηλαδή περιοχές. Αυτή η απώλεια βιοπικιλότητας που έχει γνωστές αρνητικές επιπτώσεις. Επίσης βλέπουμε, λόγω των δασοπυρκαγιών, επίσης οδηγούν σε μια απώλεια της ε, δασικής μάζας, ε, των δασών μας. Και αυτό έχει σημαντικότατες άμεσες επιπτώσεις όσον αφορά τις ίδιες τις κλιματικές αλλαγές. Εδώ υπάρχει η διασύνδεση. Αυτό που ήθελα να πω είναι η επίπτωση που έχουν οι δασοπυρκαγιές σε σχέση με τις ε, κλιματικές αλλαγές. Και με συγχωρείτε αν αυτό παρανοήθηκε ή εκφράστηκα με τέτοιο τρόπο να υπάρχει παρανόηση και δεν ήμουν επαρκώς σαφής. Εν πάση περιπτώσει δεν έχω κανένα πρόβλημα αν δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμη επαρκώς να ε, το επεκτείνω, να το σχολιάσω περαιτέρω. Πιο συγκεκριμένα χειροπιαστά θέματα και άλλα ζητήματα τα οποία απομένουν, διότι συνδέονται αυτά μεταξύ τους. Ο κύριος Ζέμπερ μας ανέφερε το θέμα του, της αποθήκευσης σύλληψης και, ε, συγγνώμη, της ε, σύμβασης για την προστασία από τις κλιματολογικές, κλιματικές αλλαγές. Έχει η Ισπανική Προεδρία σε σχέση με το Συμβούλιο και το, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόκληση να αντιμετωπίσει που θεωρούμε ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα που επομιζόμαστε ως Ισπανική Προεδρία, η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Έχουμε συνειδητοποιήσει τη σημασία της σπουδαιότητα αυτής της οδηγίας και πιθανόν δεν θα είναι εύκολη μια συμφωνία, διότι οι θέσεις εκκίνησης από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μπορεί να ε, ε, μην είναι οι ίδιες. Όμως παρόλα αυτά πιστεύω ότι ασκώντας σωστά τον διάλογο και όντας επαρκώς ελαστική και ευέλικτη και αν όλοι είμαστε σαφείς στους στόχους που θέλουμε να ακολουθήσουμε και αν όλοι είμαστε διατεθειμένοι να κινηθούμε μέσα σε συγκεκριμένα περιθώρια ε, τα οποία θα έχουν προκαθοριστεί μπορούν, μπορεί αυτό το έργο να καλυφθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ως προθεσμία. Και ένα άλλο από τα θέματα που είχαν τεθεί επίσης και που είχε χαρακτήρα κατά κάποιο τρόπο ας το πω έτσι πιο επίκαιρο ή πιο άμεσο σε αυτή την περίπτωση ε, αφορά την Ισπανία. Δεν θέλω με κανένα τρόπο να πιστέψετε ότι επειδή είμαι εδώ ως Προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ένωσης, ε, θέλω να υπεκφύγω ή να μην αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο αφορά αποκλειστικά την Ισπανία, όπως είναι η εφαρμογή του νόμου για τις παράκτιες περιοχές, Ντε Κώστας. Είμαι πρόθυμη να αφιερώσουμε μια συνάντηση αποκλειστικά σε αυτό το θέμα, ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε σύγχυση της Ισπανίας ως προεδρεύουσα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με ε, ανάμειξη αυτών των θεμάτων. Θα ήθελα να σας πω ότι όταν η Ισπανία, η κυβέρνηση της Ισπανίας εξεπώνησε το νομοθέτημα αυτό για τις παράκτιες περιοχές, λέει Ντε Κώστας, που έγινε το 1988, ήταν ένας προπομπός, πρωτοπόρος ε, νόμος σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό το νομοθέτημα και σήμερα εξακολουθεί να έχει λόγω του καινοτόμου χαρακτήρα που είχε το 1988 είναι ένα σημείο αναφοράς. Σήμερα οι αρχές αυτές είναι όλο και πιο θα έλεγα ε, φιλόδοξες στις απαιτήσει που θέτουν γνωρίζοντας τις κλιματικές αλλαγές και τις επιπτώσεις τους για τις παράκτιες περιοχές καθώς επίσης και την προστασία των παράκτιων περιοχών και αυτή είναι η πεμπτουσία, αυτή είναι η ουσία εδώ σε σχέση με την Επιτροπή σας. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο ήθελα να σας διαβιβάσω. Εμένω και επιμένω και ελπίζω ότι θα το κατανοήσετε σωστά. Προσφέρω τη συνεργασία μου για να επεξηγήσω την εμβέλεια και του τι συνεπάγεται αυτός ο νόμος, ξεχωρίζοντας όμως αυτό το θέμα από τις δραστηριότητες και δράσεις της, Ευρω... της Ισπανικής Προεδρίας ως Προεδρεύουσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην υπάρχει οποιαδήποτε εδώ δηλαδή παρερμηνία ότι εγώ θέλω να προστατεύσω εδώ κάποια ισπανικά συμφέροντα και όχι τα ευρωπαϊκά συμφέροντα που είναι ρόλος μου να ε, προασπίζομαι ως Προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Και ένα άλλο θέμα ήταν ο κανονισμός για τα βιοκτώνα και που ετέθη από τον κύριο Κλάς. Η Ισπανική Προεδρία από την κυρία Κλάσα ε, είπε κύριο Κλάση η Προεδρία. Θέλουμε να προαγάγουμε αυτό το στόχο και ιδιαίτερα αυτό το οποίο γίνεται από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δέσμευσή μα είναι να αφιερώσουμε τον αναγκαίο χρόνο για τη συζήτηση αυτού του θέματο στο Συμβούλιο. Να προχωρήσουμε το δυνατόν ταχύτερα σε μια συμφωνία μέσα στου κόλπου του Συμβουλίου, ακολουθώντα ένα παράλληλο, μια παράλληλη τροχιά σε σχέση με τη συζήτηση που διεξήχθη εδώ. Αυτό που θέλουμε είναι να γίνει μια, μια αξιολόγηση όσον αφορά τα θέματα και την πρόοδο που έχουν επιτευχθεί και υπάρχουν κάποια στοιχεία κλειδιά όσον αφορά το επίπεδο εφαρμογής, ε, την εμβέλεια ε, εφαρμογής, ε, τα προϊόντα από πλευράς βιοκτόμων, αυτό στο ένα τμήμα της συζήτησης, αποσαφήνιση των κριτηρίων αποκλεισμού κάποιων ουσιών για λόγους προστασίας της υγείας αλλά και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Εδώ επίσης έχουμε υγειονομικό κοινωνικό σενάριο και περιβαλλοντικό σενάριο που βλέπουμε και για θέματα ουσιών που αφορούν τα βιοκτώνα αλλά επίσης και ενεργές ουσίες ως συστατικά και όλα αυτά μπορούμε να τα εξετάσουμε επικεντρωνόμενοι σε αυτά. Πάντα εμένα και επιμένω στο μέτρο που θα σημειώνεται πρόοδο σε αυτέ τι εργασίε και από πλευρά Ευρωβουλή. Έτσι θα προχωρήσουμε και εμεί. Ζητώ συγγνώμη για την ταχύτητα με την οποία κάλυψα αυτέ τι παρεμβάσει ε, και ε, ζητώ συγγνώμη αν υπήρξε κάποια παρεμηνία. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Σε χρόνο ρεκόρ καταφέρατε, κυρία Υπουργέ, με διεξοδική κιόλας απάντηση που δώσατε. Αυτό θα, έχουμε, θα μας δώσει και την ευκαιρία να συνεχίσουμε το δεύτερο γύρο. Συνεχίζουμε με τις ερωτήσεις. Ραβίτε Κουνάιτε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση των προτάσεων αυτών. Οι κλιματικές αλλαγές είναι ένα σημαντικό θέμα, σημαντικό και για μας και βλέπουμε ότι υπάρχει εδώ και το ζήτημα των, της συζήτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι προπομπώς η, η Ισπανία στην αιωλική και την ηλιακή ενέργεια. Σε άλλους τομείς όμως υπάρχει ανάγκη να καλυφθεί το κενό πόρο απέχουμε από την κάλυψη του στόχου του 20%. Σε πολλά κράτη-μέλη δεν υπάρχει καν πολιτική βούληση ώστε να προαχθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δεν δραστηριοποιούνται πολλά κράτη-μέλη. Ερώτησή μου λοιπόν, η Ισπανική Προεδρία, προς την Ισπανική Προεδρία. Κάποια συγκεκριμένα μέτρα έχετε υπόψη σας ώστε να δώσετε κίνητρα στα υπόλοιπα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν με πιο ενεργό τρόπο αυτούς τους στόχους. Και Ποια είναι η αξιολόγηση, η κλιματική αξιολόγηση. Είχαμε μια οδηγία όσον αφορά τον τομέα. Σήμερα όμως δεν πρόκειται για ανεξάρτητες ε, μελέτες ε, και γι' αυτό πολλές φορές αντιμετωπίζουμε την κατάσταση ότι τα κριτήρια που από πλευράς ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υλοποιηθούν σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι προκατηλημένοι που υποβάλλουν με βάση, ας το πω έτσι, στοιχεία τα οποία δεν είναι αξιόπιστα και ε, θέλουν να επηρεάσουν τις αποφάσεις. Παράδειγμα για τον, ε, την περιοχή της Βαλτικής θάλασσας ε, και για προγράμματα τα οποία αφορούν περιοχές Natura 2000 και βλέπουμε εδώ στα ενεργειακά προγράμματα βλέπουμε να απουσιάζουν οι μελέτες επιπτώσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πώς εσείς ε, κρίνετε αυτή την ε, αμοιβαία συνάρτηση. Ευχαριστώ κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ και την κυρία Υπουργό για την παρουσία της. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνω πόσο δεσμευμένη είναι η Ισπανία σε θέματα προστασίας του εδάφους και της Λευκής Βίβλου για την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. Αυτό για άλλη μια φορά επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η προστασία του εδάφους για να προλάβουμε και τη διάβρωση του εδάφους αλλά και τις πλημμύρες αλλά και για να παρατείνουν μάλλον συγγνώμη, για την παράταση των περιόδων ε, ξηρασίας να μπορέσουμε να ε, προστατεύσουμε τα δάση μας ε, μειώνοντας τις δασοπυρκαγιές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για την Κοπενχάγη είναι σαφές ότι συμφωνώ απολύτως ότι η παγκόσμια αλλαγή του κλίματος είναι ένα πολύ σοβαρό φαινόμενο που οφείλεται και στην ανθρώπινη δραστηριότητα και θα πρέπει να έχουμε και μία επιθετική διπλωματία στο θέμα του κλίματος για να μπορέσουμε να θέσουμε και σε εφαρμογή τα ε, βασικά συμπεράσματα ε, του Μπαλί, δηλαδή αυτή την κοινή αν και διαφοροποιημένη ευθύνη. Ε, νομίζω ότι δεν παρουσιάστηκαν στην Κοπενχάγη προτάσεις οι οποίες να είναι επαρκείς προκειμένου να καταλήξουμε σε αυτό το στόχο. Αν θέλετε, είναι δύο τα φαινόμενα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατά κάποιο τρόπο. Πρώτον, να μην επιτρέψουμε στην Κίνα να κρύβεται πίσω από τις αναπτυσσόμενες χώρες και αφετέρου να υπάρχει και μία εκστρατεία για να πείσουμε τις Ηνωμένε Πολιτείες να δεχθούν ε, κάποια όρια τα οποία θα είναι και νομικώς δεσμευτικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Περέγιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες αμφιβολίε που είχαμε τις διασκεδάσατε ήδη στην παρέμβασή σα, αλλά δεν θα ήθελα να χαθεί η ευκαιρία να κάνω δύο παρατηρήσεις. Όντως ε, θα πρέπει να χαιρόμαστε όλοι για το σημείο που μα διάβασε υπουργό από πλευράς ε, Κορεπέρ, αλλά αυτά τα συγχαρητήρια δεν θα πρέπει να μας χαλαρώσουν. Είναι αλήθεια ότι έχουμε μία και μόνη θέση για το θέμα της αλλαγής του κλίματος, αλλά ορισμένες φορές συγχαίνουμε τη μία θέση με τη μία φωνή, διότι κάποιες φορές δεν μιλάμε με μία φωνή. Τι εννοώ για να γίνω πιο κατανοητές. Ναι, μεν έχουμε μία φωνή, αλλά η απόϊχοι και οι εγωισμοί ορισμένες φορές ακούγονται περισσότερο από τη φωνή μας. Ε, εάν θέλουμε λοιπόν να φτάσουμε στο Μεξικό το 2010 θα πρέπει να μιλάμε όντως με μια φωνή για να μην μας λαμβάνουν ως μια διαφοροποιημένη θέση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι μεν μας χαροποιεί το σημείωμα που μας διαβάσετε από την Κορεπέρα αλλά δεν θα πρέπει να χαλαρώσουμε και να συνεχίσουμε τις εργασίες μας μέχρι την, ε, το Μεξικό ε, και να φτάσουμε εκεί και με μια θέση αλλά και με μια φωνή. Ε, μίλησατε για το νερό, εξηγήσατε πάρα πολλά πράγματα και με αυτά συμφωνώ, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και αυτά που πρέπει να κάνουμε με τη Μεσόγειο, με τις αλλαγές του κλίματος, με τις ε, τεράστιες περιόδους ξηρασίας που βιώνουμε. Είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να αναζητήσει απαντήσεις η Ισπανική Προεδρία, τις ανακοινώσετε, αλλά αυτό θα πρέπει να ε, αποτελήσει ε, τμήμα του διαλόγου, όπως και το θέμα για τα δάση μεταξύ Βορρά και Νότου της Μεσογείου, διότι ορισμένες φορές συναντιόμαστε και μιλάμε με χαρά, με μεγάλη διάθεση, αλλά αγνοούμε ότι για να έχουμε αλληλεγγύη θα πρέπει να εργαστούμε πάρα πολύ σκληρά. Ε, να υπάρχουν μεν λύσεις από πλευρά Ισπανικής Προεδρίας, διότι εσείς είστε αυτοί που αναλαμβάνατε μετά από την πρώτη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας ε, τα ενία και θα πρέπει να προσπαθήσετε λοιπόν να υπάρχει αλληλεγγύη στο διάλογο μεταξύ Βόρεια και Νότου της Μεσογείου. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω εδώ την Υπουργό. Και να πω ότι αν και είμαι σε άλλο πολιτικό κόμμα στην Ισπανία, πιστεύω ότι πρέπει να συνεργαστούμε και εδώ είναι η μεγάλη ευκαιρία να συνεργαστούμε για τη Μεσόγειο και για μία λογική που συνήθως δεν ε, αντιμετωπίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είμαι σχεδόν 10 χρόνια εδώ και θεωρώ ότι εξακολουθεί να είναι απαραίτητο ο, προεδρίες όπως η Ισπανική να μας εξηγούν λίγο καλύτερα ποια είναι τα προβλήματα του Νότου. Προβλήματα τα οποία είναι τελείως διαφορετικά ε, στην ερμηνεία τους. Παραδείγματο χάρη το θέμα της απερίμωσης, ε, το οποίο συζητάνε μεν η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά χρόνια, αλλά δεν έχει λάβει κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση του. Ε, ε θέματα που αφορούν το παραγωγικό σύστημα και πολλά άλλα. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την κυρία Υπουργό να προσπαθήσει και θα τύχει και όλες μας τη στήριξη, τουλάχιστον τη δική μας, να προσδώσει μια κάποια γνώση, μια παιδεία για τη Μεσόγειο. Έχουμε μια γενική διευθύντρια η οποία ασχολήθηκε με θέματα έρευνας και εδώ είναι μεγάλη τύχη αυτό για μας διότι η έρευνα είναι κάτι το οποίο θα ε, συμπεριληφθεί. Ε, στις πολιτικές μας. Οι γνώσεις για τη Μεσόγειο δεν έχουν φτάσει ακόμα στην Ευρώπη και οι πολιτικές, ε, οι τουλάχιστον οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει να γίνονται και από αυτή την οπτική γωνία. Θα ήθελα να σας κάνω και μία ερώτηση. Εγώ θεωρώ ότι η συστημική πολιτική θα πρέπει να έχει μια συστημική προσέγγιση στην αλλαγή του κλίματος και την προσαρμογή. Και θεωρώ ότι οι στρατηγικές για το έδαφος είναι υψής της σημασίας δεν ε, ε, πρέπει να στεκόμαστε στο κατασκευάζω, δεν κατασκευάζω, είναι ιδιοκτησία μου ή δεν είναι ιδιοκτησία μου, αλλά στο να υπάρχει μια στρατηγική για την γεωργία, να λάβουμε υπόψη μας την αλλαγή του κλίματος, την προστασία του εδάφους, την ε, λειψιδρία, διότι, ε, το διοξίδιο του άνθρακα, διότι όλα αυτά αποτελούν ένα συνολικό πακέτο για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχει μια συνολική κατευθυντήρια γραμμή, διότι εδώ, για παράδειγμα, δεν υπάρχει συνειδητοποίηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το τι γίνεται με τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, ε, τη νομιμότητα ή μη νομιμότητα για τα θέματα του νερού. Τελειώνω σε ένα λεπτά, κύριε Πρόεδρε πρέπει να υπάρξουν νέες ιδέες και νέες μέθοδοι για μια παραγωγική αναδάσωση που ταυτόχρονα θα δεσμεύει και διοξίδιο του άνθρακα, όπως επίσης και πολλά άλλα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, είναι χαρά μας να βρίσκεστε εδώ. Στη διάρκεια της παρέμβασής σας και σε κάποιες ερωτήσεις ακούσαμε το θέμα της προστασίας των δασών. Θα ήθελα να γνωρίζω πιο συγκεκριμένα πώς η Ισπανική Προεδρία θα λάβει υπόψη τα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια αυτής της δασικής δραστηριότητας και σε αυτές τις πολιτικές προστασίες, αν θα μπορέσετε να μας δώσετε και κάποια συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία ή δυνατόν. Η Εντίτε Στρέλα. ευχαριστώ πολύ. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου και τα συγχαρητήρια για το φιλόδοξο πρόγραμμα που μας παρουσιάζεται και για την συνολική σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά τις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας. Πράγματι όλα αλληλοσυνδέονται και αλληλοσυναρτώνται. Η αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία των εδαφών και όλα αυτά συσχετίζονται με την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και την καταπολέμηση των θεομηνιών και τις θεομηνίες. Όπως είναι γνωστό, οι φυσικές καταστροφές, οι θεομηνίες είναι όλο και πιο συχνές και όλο και πιο καταστροφικές. Η ίδια η Υπουργός αναφέρθηκε και είπε ότι υπάρχουν περίοδοι πλημμυρών λόγω έντονων βροχοπτώσεων που εναλλάσσονται με περιόδους λειψιδρίας και ξηρασίας απόλυτης ξηρασίας και ότι στην ίδια περιοχή και περιφέρεια έχουμε τη μία περίοδο πλημμύρες, την άλλη φορά ξηρασία και πυρκαγιές. Τώρα, στο πακέτο μέτρων για την ενέργεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συναφή θέματα αξιολογείται ο στόχος της ενεργειακής απόδοσης και καθώς επίσης και η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε από την άλλη πλευρά τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου για την ξηρασία και τη λειψίδρια, λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη διασύνδεση θεμάτων. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια μέτρα συγκεκριμένα χειροπιαστά έχει υπόψη να υλοποιήσει και να δρομολογήσει η Ισπανική Προεδρία, ώστε να προβλέψει και να προνοήσει για να αντιμετωπιστούν οι θεομηνίες και φυσικές καταστροφές πλημμύρες, λειψιδρία, ξηρασία και δασοπυρκαγιές και που έχουν και περιβαλλοντική συνιστόσα και οικονομική και ε, κοινωνική επίπτωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σλούτερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και βλέπω ότι η Ισπανία σταμάτησε να αυξάνει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος ε, σε μεγάλο βαθμό λόγω ακριβώς ε, της πολιτικής σας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για τους φόρους στον τομέα της ε, ενέργειας. Όμως ποιοι είναι οι στόχοι σας και ποιες είναι οι πρωτοβουλίες της Προεδρίας για να μπορέσουμε να φτάσουμε τους στόχους του Κιώτο πριν φτάσουμε στο Μεξικό για την εσωτερική ε, παραγωγή σε επίπεδο κρατών μελών και επίση για την ε, μεταφορά ζωών περιμένουμε μια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει καθυστερήσει. Ε, τι κάνει η Προεδρία για αυτό το θέμα, ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, κάνει μια, να υποβάλει μια πρόταση για τη μεταφορά ζώων και ούτως ώστε να βρούμε μια λύση για καλύτερες συνθήκες μεταφοράς για τα ζώα και μέγιστο χρόνο μεταφοράς 8 ώρες. Ευχαριστώ. Και τελευταία ερώτηση από την Ισπανία και πάλι, Πιλάρα Γιούζο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη γιατί λίγο πολύ τα ρωτήσαμε όλα και τα είπαμε όλα. Ε, καλή επιτυχία στα όσα μας παρουσιάσατε. Αναφερθήκατε στο ριτς και στα χημικά προϊόντα και η κυρία Κλάς ε, σας έθεσε το θέμα των επιπτώσεων. Νομίζω ότι το Συμβούλιο θα έπρεπε να ε, προτείνει μία ε, μελέτη περιβαλλοντικών υποπτώσεων για αυτές τις δύο οδηγίες, διότι έχουμε απαγορεύσει μία σειρά από ουσίες, άρα εισαγάγουμε προϊόντα τα οποία τις χρησιμοποιούν. Και επίσης η Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου δεν θα μας επιτρέψει να μην τα εισάγουμε. Όσες επιθεωρήσεις και έλεγχοι να γίνονται σε τρίτες χώρες δεν θα γίνεται να απογορευτεί και δεν θα γίνεται να σταματήσει η εισαγωγή των προϊόντων αυτών από τρίτες χώρες. Πρέπει να γίνει λοιπόν μια αξιολόγηση αντικτύπου και θα πρέπει να την προτείνει το Συμβούλιο. Και επίσης, ε, αναφερθήκατε στην προστασία των δασών. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να μιλάμε και ε, για την ε, δημιουργία δασών. Νομίζω ότι είναι ένα ακόμα μέτρο για να ε, αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματος, ένας ακόμα τρόπος για να δεσμεύουμε διοξίδιο του άνθρακα και να, τον, ε, να το αποθηκεύουμε. Μιλήσατε και για κοινή αγροτική πολιτική. Στην Επιτροπή Γεωργίας εγκρίθηκε μια έκθεση η οποία ζητά συγκεκριμένα να γίνει μια ευρωπαϊκή δασική πολιτική. Εσείς δεν θεωρείτε ότι είναι κάτι τέτοιο απαραίτητο. Θα κάνετε κάτι για να προωθήσετε μία αποκλειστικά ευρωπαϊκή δασική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κλείνει και ο δεύτερος γύρος των ερωτήσεων. Τώρα έχουν μείνει περίπου 10 λεπτά και δίνουμε το λόγο στον Υπουργό για να απαντήσει. Προσπαθήσω πραγματικά να προσαρμοστώ στο χρόνο αυτών των 10 λεπτών στις απαντήσεις μου. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ένα από τα θέματα που έθεσε ε, η Ευρωβουλευτής είναι τα θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Λοιπόν, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπάρχει νομίζω μια πολιτική βούληση από πλευρά της Ευρώπης ε, να επιτύχουμε την ε, ε, ολοκλήρωση του στόχου του 20% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2020. Η πορεία που ακολουθήθηκε από κάθε ένα από τα κράτη-μέλη είναι διαφορετική. Και εδώ πάλι πρέπει να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε και να δούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες πηγές ενέργειας που μπορούν να συνδέονται περισσότερο με την γεωγραφική θέση ενός κράτους μέλους και σαν συνέπεια αυτού να έχουμε ας πούμε κάποιους, μέσους, ε, κάποιους πόρους, φυσικούς πόρους ε, που μπορούν να ευνοούνται και άλλοι όχι. Δεν μπορούμε πολλές φορές να κάνουμε λόγο για την εκμετάλλευση, για παράδειγμα, ηλιακής ενέργειας ε, με ισότιμη αντιμετώπιση ηλιοφάνειας όταν κάνουμε λόγο για μια μεσογειακή χώρα και όταν κάνουμε λόγο για μια χώρα στη Βόρεια Ευρώπη. Αυτή η αντιστάθμιση μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα για παράδειγμα σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης με την αιωλική ενέργεια για παράδειγμα σε σχέση με άλλη χώρα που βρίσκεται στη Μεσόγειο. Εγώ αυτό που θα κάνω είναι θα προσπαθήσω να διαβιβάσω το μήνυμα αυτού που είπατε και να συμμεριστούμε και να επιμερίσουμε ενέργειες και πληροφορίες ε, ενεργειακά και ενημερωτικά και έτσι με αυτόν τον τρόπο να συνενώσουμε προσπάθειες ώστε να πετύχουμε αυτό το στόχο που νομίζω ότι και εσείς συμμερίζεστε πλήρως και αυτά που διαβιβάζονται εδώ είναι οι μεγάλες ανησυχίες σας και τα κυριότερα μελήματά σας. Επίσης έγινε αναφορά σε εκείνο που ήταν σε αυτό που είναι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρέπει μεταξύ μας να προσπαθήσουμε κυρίως οι διατάξεις που έχουμε να έχουν μια σωστή εφαρμογή, αποτελεσματική εφαρμογή. Η νομοθεσία που εφαρμόζεται πρέπει να εφαρμόζεται σωστά και αποτελεσματικά. Και έτσι είναι αυτονόητο φυσικά ότι οι κοινοτικέ διατάξεις συνεπάγονται μια έντονη σε βάθο ε, συμμετοχή του δημοσίου και ε, όλων στην ε, προσπάθεια αυτή και επιπλέον να διασφαλίσετε η διαφάνεια. Να μην σκεφτόμαστε μόνο ποιο ε, εκπονεί μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά η διαδικασία ενημέρωση ε, πρέπει εκεί να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Και έτσι λοιπόν σε σχέση με περιπτώσει όσον αφορά τη δημόσια ενημέρωση και πληροφόρηση θα πρέπει προβλήματα που ίσω υπάρχουν να επιληθούν με τον πιο θετικό τρόπο. Επιπλέον ένα επιπρόσθετο θέμα. Κάνουμε λόγο εδώ για μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια και ότι ιδιαίτερα ως προς αυτό πορευόμαστε πιο πέρα από τον ίδιο τον περιορισμένο ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό θέλω να το συνενώσω με το θέμα της διαφάνειας. Να μην σκεφτόμαστε ότι επειδή μια χώρα είναι όμορη χώρα με μια άλλη και με μια χώρα που μπορεί να μην είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς ε, ε, ε, δεν θα πρέπει να υλοποιούμε τις προδιαγραφές για τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να μην σεβόμαστε αυτές τις πτυχές. Υπάρχουν κράτη-μέλη και εδώ προσφέρομαι ιδιαίτερα για να σας διαθέσω τα αντίστοιχα στοιχεία που στην ιστοσελίδα web που έχουν από πλευράς ε, των στοιχείων και ε, στην ιστοσελίδα εμπεριέχονται τα στοιχεία για παράδειγμα περιβαλλοντικών επιπτώσεων ώστε οποιοδήποτε πολίτης έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ να μπορεί να συμβουλευτεί αυτά τα, τα στοιχεία από την ιστοσελίδα. Σας το λέω αυτό, υπάρχει αυτό το θέμα και θα ήθελα να το πω στους ευρωβουλευτές ε, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε, να προχωρήσουμε ως προς αυτό το στόχο. Ο κύριος Πρόντι μας έκανε λόγο για τα εδάφη και την προστασία τους ε, και εδώ για την πρόθεση να ε, υπάρξει προσπάθεια διασφάλισης των εδαφών. Μας έκανε λόγο επίσης για τη λειψιδρία και την περιόδους ξηρασίας. Εδώ θα ήθελα να γίνει κατανοητό πώς μπορούμε να εργαστούμε, πώς το βλέπω εγώ. Αν έχουμε μία περίοδο ξηρασίας, η δική μας ε, άποψη και προσέγγιση είναι η Ευρώπη να έχει ένα στρατηγικό πρόγραμμα, ένα σχέδιο Τώρα ο τίτλος ε, σε σχέση με αυτό πρέπει να μπορεί να έχει τέτοια μορφή ώστε να αντιμετωπίζεται γενικά αυτή η ξηρασία με τέτοιο τρόπο ώστε κανένας ευρωπαϊκής, ε, ευρωπαίος πολίτης να μην στερείται το νερό. Όμως παράλληλα καθώς θα εργαζόμαστε για όλες τις πολιτικές που μπορούμε να δρομολογήσουμε και να καταστήσουμε αποτελεσματικές ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιες ε, περιπτώσεις ξηρασίας ή τουλάχιστον να ε, σημειώνονται με μικρότερη συχνότητα από ό,τι μέχρι σήμερα. Εδώ λοιπόν είναι αυτονόητο ότι ό,τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών είναι το καλύτερο εργαλείο, το καλύτερο μέσο που έχουμε στα χέρια μας ε, για τις διαδικασίες αυτές για τη διαφύλαξη των υδάτινων πόρων. Και συμπίπτω απόλυτα στην άποψη αυτή μαζί σας και ότι σε σχέση με την πρώτη μου παρέμβαση όσον αφορά τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε, ε, έκανα λόγο για τις αναδυόμενες χώρες, για τις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά εδώ επιμένω και εμένω ότι η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών είναι παγκόσμια, είναι συνολική και σφαιρική και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά τα οποία λέτε. Όμως στην Ευρώπη πρέπει να συνεχίσουμε να προχωράμε με αυτά τα θέματα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κάποιοι να κατέβουν από αυτό το τρένο, να αποβιβαστούν και να μην συμμετέχουν σε αυτή την κοινή πορεία. Το αντίθετο. Εμείς είμαστε πρωτοπόροι στο παρελθόν στην Ευρώπη. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε πρωτοπόροι. Όχι μόνο πρωτοπόροι, αλλά και εκείνοι οι οποίοι μέσα σε αυτό το μεγάλο διεθνές πλαίσιο θα μπορέσουμε να ε, πετύχουμε μια κοινή δράση στο Μεξικό να ε, ενώσουμε τις προσπάθειές μας για μια κοινή δράση όλοι και σε σχέση με αυτό το οποίο είπε ο ε, άλλος Ευρωβουλευτής ε, και συμπίπτω μαζί του στην άποψή του ότι πολλές φορές ε, για το να μιλάμε με μία ενιαία φωνή υπάρχουν πολλές φορές προσωπικά συμφέροντα και ιδιοτέλεια παρά μία ενιαία ενωμένη φωνή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεσμεύομαι από πλευρά τη Ισπανική Προεδρία να διαβιβάζουμε κοινά μηνύματα με ενιαία φωνή από πλευρά μα. Να εμπλουτίζονται αυτά τα κοινά μα μηνύματα από όλους μας και αυτό νομίζω μπορεί να είναι ένα εγχείρημα συνένεσης με αυτή την Ευρωβουλή από πλευράς μας και πάντα να προσπαθούμε να προχωρούμε έστω και με πολύ μικρά βήματα αλλά με βήματα μικρά αλλά ασφαλή ώστε να διασφαλίσετε η ενότητα της, Ευρω... της έκφρασης της Ευρώπης για τα μέτρα καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Το ίδιο και στο διεθνές, στο παγκόσμιο επίπεδο και με ένα στόχο πολύ σαφή και με ε, μια ημερομηνία που πρέπει να είναι εφέτος 2010 στο Μεξικό ημερομηνία και τοποθεσία. Ένα άλλο θέμα ήταν η έλλειψη, η Ισπανίδα των υδάτινων πόρων του νερού και ιδιαίτερα στο τόξο της Μεσογείου, στη Νότια Ευρώπη. Εδώ επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω κάτι. Το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια κοινοποίηση, μια ανακοίνωση για την σπανίδα του νερού και τη ξηρασία με μια σειρά πολιτικών προτάσεων, πολιτικών ε, για, που πρέπει να ακολουθηθούν σε εθνικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο και ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπιστεί η λειψιδρία και η σπανίδα των υδάτινων πόρων. Τότε είχε λεχθεί ότι θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια ομάδα πραγματογνωμόνων αξιωματούχων υπό την Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που συνεισέφερε με μια σειρά συστάσεων για τα προγράμματα διαχείρισης ε, του νερού και τα συναφή. Υπό την Ισπανική Προεδρία βέβαια τώρα και έχοντας συνειδητοποιήσει ότι η Μεσογειακή περιοχή, η Μεσόγειος έχει ιδιαίτερα ξεχωριστά χαρακτηριστικά στοιχεία, θέλουμε τελεσίδικα και καθοριστικά να προαγάγουμε την λήψη αποφάσεων και την επίτευξη μιας ευρωπαϊκής τελικά στρατηγικής που θα μειώνει τις κοινωνικές επιπτώσεις, τις κοινωνικές επιπτώσεις και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την αύξηση των ε, ε, περιπτώσεων ξηρασίας στην Ευρώπη και ιδιαίτερα να ληφθεί υπόψη η περιοχή της Μεσογείου. Υπάρχουν δύο σύνοδοι, δύο σκέψεις ε, που έκανα αναφορά στην παρέμβασή μου που θα μας βοηθήσουν να εμπλουτίσουμε αυτές τις δράσεις μας. Η κυρία Γκουτιέρε τώρα στη συνέχεια μα έκανε λόγο για την ανάγκη έρευνας και φυσικά είναι απαραίτητο αυτό το στοιχείο. Το είπα ήδη στην πρώτη μου παρέμβαση όταν έκανα λόγο για την αποθήκευση του άνθρακα, σύλληψη και αποθήκευση του άνθρακα. Οποιαδήποτε από τις ε, δραστηριότητες αυτές, ε, σε οποιαδήποτε από αυτές τις δραστηριότητες αναφερόμαστε και όταν κάνουμε λόγο για το μέλλον και το περιβάλλον πρέπει χέρι με χέρι να αναπτύσσονται αυτές ε, οι ερευνητικές δραστηριότητες. Είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω χθε σε μια σύσκεψη, σε μια διάσκεψη στην Ισπανία για θέματα βιοπικιλότητας ακριβώς. Και νομίζω ότι συνδέεται η χθεσινή ημερίδα με αυτά τα οποία αναφέρθηκαν εδώ και είπατε κι εσείς για τη δημιουργία μιας διεθνούς πλατφόρμας για θέματα βιοπικιλότητας για να ακολουθηθεί παράλληλη πορεία από πλευρά των προσπαθειών μας. Είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για αυτά τα οποία αναφέρατε. Για τα θέματα γεωργίας ξεπέρασα τον χρόνο που μου δώσατε πρόεδρε τα 10 λεπτά. Όμως εισαγάγαμε και θα έχω ευκαιρία και από πλευρά Επιτροπής Γεωργίας ε, του Ευρωκοινοβουλίου απόψε σήμερα το απόγευμα να τα εκθέσω αυτά. Εισαγάγαμε το θέμα των κλιματικών αλλαγών επίσης ε, και επίσης ε, εισαγάγαμε και το θέμα της καταπολέμησης όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές στο περιβάλλον και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων και την αντιμετώπιση τους. Επιτρέψτε μου τώρα να είμαι πιο σύντομη και να πάω ταχύτερα, αλλά θα έχω και θα έχετε εσείς φυσικά το απόγευμα να γνωρίζετε αυτές τις θέσεις μας σε μεγαλύτερο βάθος, πιο εξειδικευμένα. Το θέμα των μεταφορών ζών των ζώων που ανέφερε ο κύριος Σλούτερ. Εδώ έχουμε διαφορετικά θέματα τα οποία συσχετίζονται με ζώα και με τη μεταφορά ζώων και την προστασία των ζώων αυτών. Αφενός έχουμε τα ζώα, τα εικόσιτα ζώα, ζώα συντροφιάς, που πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία το δυνατόν πιο σύντομα ώστε να μπορέσει να, να ισχύσει ένας νέος κανονισμός τον Ιούλιο. Από την άλλη πλευρά έχουμε την πρόταση οδηγίας για την ευεξία ευημερία των ζώων αλλά και για ζώα που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς ε, σκοπούς για την έρευνα. Και υπάρχει νομίζω πολιτική συνένεση από πλευράς του Κοινοβουλίου για τα τεχνικά τμήματα αυτού του φακέλου και για τα θέματα επιτροπολογίας ε, που εκκρεμούν και που συνδέονται με την συνθήκη της Λισαβόνας. Και από την άλλη πλευρά έχουμε το θέμα της ετικετοποίησης, ε, της, ε, του, ε, της ετικετοποίησης ώστε να γνωρίζουν οι καταναλωτές τι ακριβώς γίνεται από πλευράς μας. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια ίσως και νομίζω μια παρόμοια συζήτηση διεξήχθη σήμερα εδώ για την ετικετοποίηση, έτσι δεν είναι όχι βέβαια που να αφορά την ευεξία των ζώων, για να μην υπάρχει όμως μεγαλύτερη σύγχυση, αλλά για να διευκολύνουμε τους καταναλωτές να διευκολυνθούν, να κατανοήσουν τι ακριβώς εμπεριέχει ένα προϊόν, ένα ε, ε, συγκεκριμένο προϊόν. Και έτσι επίσης και το θέμα της, ε, του προγράμματος κοινοτική δράσης για την ευεξία και ευζοία των ζώων. Είναι θέματα που είναι παράλληλα και που σε διάφορους υποτομείς, ας το πω έτσι, αναπτύσσονται και εξελίσσονται, αλλά νομίζω εκείνο το οποίο πιο γοργά μπορεί να αντιμετωπιστεί είναι η, κίνηση, η διακίνηση ζώων, η κόστη των ζώων και η ευεξία των ε, ζώων όσον αφορά την χρήση τους για επιστημονικούς σκοπούς. Και για τα περαιτέρω, μια και είναι δυνατόν ε, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας να μην ε, μπορέσει να ολοκληρωθεί ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο θα δοθεί συνέχεια στην επόμενη Προεδρία. Ζητώ συγγνώμη για το ότι κατηγοριοποιώ τώρα ε, παρεμβάσεις αυτά τα οποία αναφέρθηκαν από την κυρία Αγιούσο, την κυρία Εστρέλα και από Ευρωβουλευτή που αφορούν ένα κοινό θέμα. Πρέπει να κάνουμε, όταν κάνουμε λόγο για τα δάση, πρέπει να κάνουμε λόγο για τα δάση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, σε ένα πλαίσιο περιβαλλοντικό. Πρέπει να εντάσσονται και σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και να γίνεται και μια εξέταση αναφορά σε ένα οικονομικό πλαίσιο, οικονομική εμβέλεια. Να σκεφτούμε ότι στην Ευρώπη των 27 κρατών μελών η δασική κάλυψη είναι κάτι παραπάνω από 42%. Και αυτό το ποσοστό, αυτό ο αριθμό ω μέγεθο μπορεί να εξηγήσει αφ' το ενδιαφέρον και συμφέρον για την προστασία και διατήρηση διατήρηση και συντήρηση των δασών. Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι. Για κάποιους από αυτούς αναφέρθηκα ήδη στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, την απώλεια της βιοπικιλότητας, την ε, ε, επέκταση της ε, ερημοποίησης. Τα δάση είναι αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Είναι βιότοποι χλωρίδας και πανίδας που συνεισφέρουν στη διατήρηση και διασφάλιση της βιοπικιλότητας και διαδραματίζουν ένα ρόλο θεμελιώδου σημασία στον κύκλο των υδάτινων πόρων του νερού και στην διασφάλιση των εδαφών και δημιουργούν ένα σενάριο κοινωνικών οικονομικών δραστηριοτήτων που σε πολλές περιοχές της υπαίθρου διασφαλίζουν πόρους ε, όσον αφορά την κοινωνία και δίνουν θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία. Αυτό μας δίνει πολλούς λόγους, αυτά όλα μας δίνουν πολλούς λόγους για να διεξαχθεί μια συνδιάσκεψη στο υψηλότατο, στο ανώτατο επίπεδο για την προστασία των δασών, ώστε να διευκολυνθεί αυτή η συνένεση κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική για την προστασία των δασών. Ζητώ συγγνώμη που ξεπέρασα τον χρόνο μου. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ. Νομίζω ότι ήταν θεμελιώδη θέματα αυτά τα οποία συζητήσαμε και περιεκτικά σε μια μισή ώρα βλέπετε πόσο ενδιαφέρονται οι ευρωβουλευτές. Είδαμε όμως και πόσο ενδιαφέρεστε εσείς και τι προσπάθειες καταβάλλετε. Χαίρομαι λοιπόν και προσβλέπω στους επόμενους έξι μήνες στο εξάμεινο της Ισπανικής Προεδρίας και ελπίζουμε ότι θα στεφθεί με επιτυχία η Προεδρία σας κάθε επιτυχία σας ευχόμαστε στο Συμβούλιο. Θα συνεχίσουμε εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ που ήρθατε και ελπίζω να σας ξαναδούμε στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Λίγη συνεδρία.